Uh, Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε παρακαλώ. Πρόκειται για μια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Τέλεια. Έχετε λάβει το σχέδιο μέρης της διάταξης. Δεν βλέπω αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις. Τα διάφορα στο τέλος συνεδρίασης. Αν έχετε ανακοινώσεις, σας παραπέμπω στα διάφορα. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Σημείο 2. Η Χριστουγεννιάτικη δεξίωση, το Χριστουγεννιάτικο ποτό, ευχάριστη ανακοίνωση. Σχεδόν ολοκληρώσαμε το πρώτο εξάμεινο της νέας κοινοβουλευτικής μας θητείας. Βλέπετε πως περνάει ο καιρός, αστραπή. Μόλις 4,5 χρόνια μας έχουν απομείνει από την κοινοβουλευτική θητεία και σας ευχαριστώ θερμά και για την αγαστή συνεργασία και την πολύ καλή αφετηρία που κάναμε. Όλες οι ακροάσεις μας πήγαν λαμπρά. Οπότε δικαιούμαστε ένα χριστουγεννιάτικο ποτό. Θα σας το προσφέρουμε και στις 3 Δεκεμβρίου, γύρω στις 6 το απόγευμα. Αν καταφέρουμε μέχρι τις 6 να διεκπαιρεώσουμε το πρόγραμμα εργασιών μας, και αν είμαστε καλά οργανωμένοι και συντονισμένοι, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε το χριστουγεννιάτικο ποτό μας. Και νομίζω ότι το περιμένουμε όλοι διακάως αυτό για να συναντήσουμε και πιο ελεύθερα μεταξύ μας, αλλά και να συζητήσουμε και για το πολύ σημαντικό μέλλον που μας περιμένει. Αυτή ήταν η μόνη ανακοίνωση του Προέδρου την κράτησα ως ξεχωριστή, πολύ σημαντική, εν ώψη των Χριστουγέννων. Σημείο 3. Εφαρμογή του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Τρέχουσα κατάσταση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον εδώ και αρκετά χρόνια Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ρόπερτ Γιάν Σμιτς, που είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας. Κύριε Γενικέ, λοιπόν, θα θέλαμε να, σας να μας ενημερώσετε συντομία για την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Γιατί θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα αυτό την πενταετία που έχουμε μπροστά μας και είναι το, το σημαντικότερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από δημοσιονομική σκοπιά και πολύ σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ανάπτυξης και αύξηση των επενδύσεων. Αφορά λοιπόν και την επενδυτική μας πολιτική, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και θέλουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην εφαρμογή αυτού του περίπλοκου προγράμματος και φιλόδοξου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν για την παρουσία σας εδώ κύριε Γενικέ Διευθυντή και σας δίνω το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Πάνω κάτω. Σας ακούμε. Increasingly studies. Και καλησπέρα σε όλους. <clears throat> Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι η καινοτομία καλύπτει το 62% της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, κυρίως από το 1995 μέχρι το 2007, κατά αυτή την περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο Πρόεδρο Ιούνκερ είχε μια πολύ φιλόδοξη ημερήσια διάταξη και αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί αν ε, συνεχίσουμε και εμεί τις καινοτομίε σε περιφερειακό ε, και εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές ε, μήνυμα που ο νέος Επίτροπος Μόιντας, ο Επίτροπος για την Καινοτομία και την Έρευνα παρουσίασε σε ακρόαση σε αυτήν την Επιτροπή. Πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στην επιστήμη και στην καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πράττουμε χάρη και των δικών σας ε, προσπαθειών. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους φτάσαμε σε μια συμφωνία όσον αφορά τον ε, πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 πρικοδοτημένο με 80 δις ευρώ. Όχι τόσο όσο είχατε ζητήσει, αλλά παρόλα αυτά είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο του 7, μια αύξηση κατά 30% και μην ξεχνάμε ότι παράλληλα μειώνεται ο κοινοτικό προπολογισμό. Μέχρι το 2020 ο προπολογισμό τη Ένωση θα είναι μικρότερο από αυτό που είναι σήμερα. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον το ότι η επιστήμη και η καινοτομία ε, θα είναι μόνο τομεί με περισσότερα κονδύλια. Μιλάμε για τον ορίζοντα 2020 για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα ρήγμα με το παρελθόν, κάτι το οποίο εσείς επίμονα ζητήσατε συνδυάζουμε την επιστήμη με την καινοτομία και αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο να έρθουν κοντήλια στην αγορά, άρα δηλαδή ε, περισσότερες επιδείξεις, ε, περισσότερα προγράμματα και εστιάζουμε την προσοχή μας στη βάση, όχι τόσο στην επιστημονική πειθαρχία. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, κατέδειξε τις προτεραιότητες, ε, γύρανση πληθυσμού, ε, κυβερνοασφάλεια, πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Δίδουμε σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και εσείς μάλιστα ζητήσατε το 20% του προεπλογισμού να χορηγείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, η επιστήμη ε, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανθρωπιστικές ε, επιστήμες. Εσείς ζητήσατε ε, τον διπλασιασμό των κονδυλίων για το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο και το πράξαμε αυτό. Επίσης, ε, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει απλούστευση. Οφείλουμε να απλουστεύσουμε τους κανόνες και τις διαδικασίες. Και τέλος, οφείλουμε και είναι σημαντικό να ανοίξουμε όλα αυτά τα προγράμματα γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει ε, χάσμα ανάμεσα στο βορρά, τον νότο, την Ανταλή και τη Δύση. Α δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Χάρη της απόφασης που βρισκομαστε τωρα χαρη της αποφαση που λαβατε τον Νοέμβριο του περασμένου έτου, μπορέσαμε τον Δεκέμβριο του 2013 να παρουσιάσουμε ε, διαγωνισμό πρόσκληση ενδιαφέροντο. Και θα ήθελα να αναφέρω κάποια στατιστικά δεδομένα. Πρώτα, η πύλη μας η πύλη ενημέρωσης λαμβάνει 3 εκατομμύρια χτυπήματα κάθε μήνα. Μέχρι τώρα λοιπόν λάβαμε 35.000 προτάσεις. 60.000 εμπειρογνώμονες είναι καταχωρισμένοι στην δική μας την τράπεζα δεδομένων. Αυτό δείχνει ότι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμά μας είναι τεράστιο και οι άνθρωποι εκτιμούν ιδιαίτερα τη νέα προσέγγιση που και χάρη της δικής σας υποστήριξης μπορέσαμε να υλοποιήσουμε. Ας δούμε τώρα τι κάνουμε για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν πέρυσι. Πρώτα απ' όλα, Δίδουμε σημασία ε, στις προτεραιότητες μας ε, το εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το είχατε στην καρδιά σας και εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Παράλληλα, δρομολογούμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, για τις καινοτομίες με μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη ταχύτητα 100 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το πρόγραμμα και στις 9 Ιανουαρίου θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση. Ο κύριος Έρλαχ δέχτηκε να παραστεί και να εγγενιάσει αυτή την καινοτομία που θα είναι καινοτομία fast track με μεγάλη ταχύτητα, υλοποίησης με μεγάλη ταχύτητα. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις ανανόμενες πηγές ενέργειας, ε, στην ενεργειακή απόδοση και πολλά άλλα. Πάνω από 85% της ενέργειας προβλέπεται για αυτούς τους τομείς. Και εσείς το ζητήσατε το 85% του προπολογισμού να διατεθεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 50% προσημειώνουμε στους διαγωνισμούς για την ανάκαμψη στην αγορά και αυτό εσείς το είχατε ζητήσει, άρα δηλαδή πρέπει να γίνει και στην πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος ε, το πράξαμε. Ε, υπάρχει και το επιστημονικό ε, φόρουμ, το πάνελ για την υγεία. Εδώ υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση. Η κυρία Μαντουρέλ και η κυρία Καβάλιο, που δεν είναι όμως μέλη αυτής της Επιτροπής πια, αλλά είναι εκείνες που ζήτησαν να υπάρχει ένα επιστημονικό συμβούλιο για την υγεία. Αυτό λοιπόν το συμβούλιο συστάθηκε και θα συνεδριάσει στις 30 Ιανουαρίου για πρώτη φορά. Κατόπιν, όσον αφορά στην απλούστευση, εφαρμόζουμε πλήρως τα μέτρα απλούστευσης ε, που είχατε συμφωνήσει κι εσείς ε, για όλους τους μετέχοντες να υπάρχει ίδια τιμολόγηση, ε, να διατίθεται ταχύτερα τα κονδύλια, το VAT, ε, το ΦΠΑ με να υπολογίζεται και να προσμετράτε και επίσης Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε ένα σημαντικό βραβείο, μια διάκριση για την τον πιο φιλικό τρόπο του να συντάσει κανείς έγγραφα. Αυτή η διάκριση μας χορηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από ανεξάρτητους δημοσιογράφους και νομίζω ότι αυτό αποτελεί αναγνώριση του γεγονότος ότι τα έγγραφά μας, οι συμφωνίες χορήγησης κονδυλίων θα παρουσιάζονται με πολύ πιο φιλικό τρόπο προς το χρήστη. Άρα δηλαδή αυτά όλα δείχνουν ότι ε, παραμένουμε προσιλωμένοι στις ε, συμφωνίες. Και όσον αφορά θέματα φύλου, τη διάσταση του φύλου. Είπατε το 40% των επιτροπών που έχουμε θα πρέπει να απαρτίζονται από γυναίκες. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή θέλουμε να είμαστε πιο προχωρημένοι, να είναι 50%. Άρα δηλαδή κατά περίπτωση λάβαμε υπόψη μας αυτά που σας είναι σημαντικά και θέλουμε να τα υλοποιήσουμε. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα νομίζω ότι προχωράμε καλά. Θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο, δηλαδή Δηλαδή το Κοινοβούλιο ζήτησε επίμονα τη δυνατότητα ο δημοσιονομικός κανονισμός να προβλέπει και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για το άρθρο 125. Εμείς καταφύγαμε πρόσφατα στο άρθρο αυτό για μια έκτακτη ανάγκη για τον ιό έμπολα. 24 εκατομμύρια ευρώ ήταν το ποσό και σε δύο εβδομάδες μπορέσαμε όχι μόνο να καταθέσουμε τις προτάσεις αλλά να γίνει και αξιολόγηση και η ε, εμβολιασμό θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Προχωρήσαμε λοιπόν γρήγορα λόγω του ότι υπήρχε αυτό το εργαλείο στο δημοσιονομικό κανονισμό. Τώρα, λίγα λόγια για το ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Γιατί ξέρετε, πράγματι προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στη συμφωνία μας, αλλά υπάρχουν και απρόβλεπτες προκλήσεις. Και αυτή που είναι η μεγαλύτερη για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πάρα πολλές υπερβολικές προτάσεις. Αν σας αναφέρω ε, ότι πήραμε ας πούμε 35.000 προτάσεις, δεν έχουμε κονδύλια για να καλύψουμε έστω και τις καλές εξ αυτών. Το ποσοστό ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ χαμηλό και αυτό είναι απογοητευτικό σε ορισμένους τομείς ε, το ποσοστό της επιτυχίας είναι μία πρόταση στις 10. Ε, σε άλλους τομείς μία στις 8. Ε, στο ιατρικό πρόγραμμα το ποσοστό επιτυχίας είναι ένα, μία πρόταση στις 30. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα, αλλά και εσείς ήσασταν ιδιαίτερα σοφοί όταν προτείνατε τα 100 δις για το ορίζοντας 2020. Θα έπρεπε να σας ακούσει το Συμβούλιο και όχι να πει 80. Έχουμε λοιπόν έλλειψη κονδυλίων και υπερβολικές προτάσεις που κατατίθενται σε εμά. Η δεύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών. Σας το είχαμε ήδη πει αυτό και στην Επιτροπή σας του Προϋπολογισμού το Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια άρχισε να κάνει περικοπές στις πιστώσεις πληρωμών και αυτό μας ανάγκασε να περιορίσουμε την προχρηματοδότηση και να αναβάλουμε διαγωνισμούς. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό και να αγοράζουν εξοπλισμό. Όταν ξεκινάει κανείς ένα ερευνητικό πρόγραμμα αμέσως χρειάζεται ρευστά για να προχωρήσει. Αναγκαστήκαμε να ε, περικόψουμε τις προκαταβολές και αναβλήθηκαν προγράμματα λόγω αυτού. Εφέτος κάπως τα καταφέρνουμε, αλλά του χρόνου θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και έχουμε υπολογίσει ότι αν αυτή η τάση της, ε, της περικοπής ε, των πιστώσεων πλεμών συνεχιστεί ε, μέχρι το τέλος του 2020, τότε το 40% των υποχρεώσεών μας δεν θα καλυφθούν από πληρωμές και αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε και ευχαριστούμε που έχουμε την υποστήριξή σας. Υπήρξε πριν από το καλοκαίρι μια συζήτηση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο και εκεί η Επίτροπος παρενέβη και είπε ποιες θα ήταν οι συνέπειες ε, πάρα πολλά προγράμματα δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν και πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να στηριχτούν. Και νομίζω ότι τελικά δεν το καταρτήσαμε αυτό το πρόγραμμα για να το υπονομεύσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη πρόκλησή μας, δηλαδή η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών. Δεύτερη πρόκληση, ε, το θέμα των κοινωνικών επιστημών και ανθρωπιστικών επιστημών, την πλήρη ένταξή του στα προγράμματά μας. Δεν μπορέσαμε ακόμα αυτή τη διάσταση να την εντάξουμε στα περισσότερα προγράμματα. Και τι εννοώ, όταν ε, ξεκινάει μία πρόσκληση ενδιαφέροντα, πούμε για το Alzheimer. Δεν πρόκειται για ένα ιατρικό και μόνο θέμα. Είναι απαραίτητο να λάβει χώρα και ερευνητικό πρόγραμμα, συνέπειες για την κοινωνία, θέματα οργάνωσης. Εάν και εκατομμύρια ανθρώπων ασθενήσουν, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην οργάνωση της κοινωνία. Είναι λοιπόν σημαντικό οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα από κοινού με τους γιατρούς. Εκεί λοιπόν δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Και τέλος, εξίσου σημαντικό, ένας τομέας που μας απασχολεί ακόμα είναι το θέμα της διεύρυνσης. Η καινοτομία διαιρεί και η επιστήμη ε, όμως δεν πρέπει να περιζόμαστε. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία για να βοηθήσουμε τις περιοχές εκείνες που δεν έχουν ακόμα τη βάση για την καινοτομία για να κάνουν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αριστείας. Και έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε τα απαραίτητα κονδύλια για την ευφυή εξειδίκευση για να βοηθηθούν οι περιοχές και οι χώρες που ακόμα δεν έχουν ισχυρή επιστήμη, επιστημονική βάση για να μπορούν και αυτές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Σε 12 περίπου λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Όπως είπατε κύριε Γενικέ, τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας είναι από τους ε, προϋπολογισμούς ε, που διασφαλίστηκαν και χαίρομαι που έχουμε εδώ τον, ε, τον πρώην Επίτροπο Προϋπολογισμού, τον κύριο, τον κύριο Λεβαντόφσκι. Βέβαια, στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε και τους αιτήσεις προϋπολογισμούς, γιατί για του χρόνου το Συμβούλιο πρότεινε περικοπές μέχρι και 10% και από τις πιο υψηλές ήταν στο τομέα μας, στην έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε πυγμή και στο μέλλον για να διαφυλάξουμε αυτό το προπολογισμό. Και εδώ μιλώ για την πρόταση του Συμβουλίου. Δεν ήταν πρόταση ρήκνωση ή πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε τώρα στη συζήτηση. Μόνο έναν εισηγητή έχουμε. Ένα αλλά σημαντικό από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Τον κύριο Κρίστιαν Έλερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή που ήρθε. Όπως είπε και ο πρόεδρος, θα, έχουμε μια, θα δημιουργήσουμε μια μόνιμη επιτροπή για τον ορίζοντα 2020 και θα κάνουμε μια ενημέρωση για τα πρώτα διδάγματα που αντλήσαμε από την εφαρμογή του. Εγώ πάντως θα ήθελα τις πληροφορίες που δώσετε στο Συμβούλιο για τα διδάγματα που αντλήθηκαν ε, αυτόματα να, τα, να τις διαβιβάζετε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί προσπαθούμε τώρα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και ένα πρώτο απολογισμό. Σε ό,τι αφορά τα βασικά ζητήματα του προϋπολογισμού, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας και νομίζω ότι είναι ακόμη πιο τραγικά τα πράγματα αν τα συγκρίνουμε με το πρόγραμμα εργασιών για το 2014-2015. Έχαμε 15 δις και είχαμε μετά για 9,3 δις το 2014 και το 2015 θα πέσουμε και κάτω από το όριο του ερευνητικού προγράμματος πλαισίου 7, του προηγούμενου. Αυτό είναι άνευ προηγουμένο. Και πέραν της σπουδαιότητας της καινοτομίας, πολύ σημαντικό θέμα είναι εδώ, ότι δεν τηρούμε μία ε, λογική και σταθερή γραμμή στην προκήρυξη των διαγωνισμών. Και οι ενδιαφερόμενοι πραγματικά διαρωτούνται αν αξίζει τον κόπο να εμπλακούν σε τέτοια προγράμματα με κοινοτικά κονδύλια. Γιατί δεν είναι σαφέ ότι θα εξασφαλιστούν τέτοια κονδύλια και στο μέλλον με τη συρρήκρωση τη διαδοχική. Επιπλέον, βλέποντας αυτή την τεράστια υπερπροσφορά και τον καταιγισμό με προτάσεις, ε, πού οφείλεται, έχουμε μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ε, μεγαλύτερους ομίλους που ενδιαφέρονται σε ό,τι αφορά το ποιοι δηλώνει υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς ε, μας ενδιαφέρουν πιο λεπτομεριακά στοιχεία για να δούμε πού οφείλεται αυτή η υπερπροσφορά. Γιατί είπατε ότι πάνω από τις μισές προτάσεις δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν λόγω της ε, οικονομικής δυσπραγίας των προβλημάτων στον προπολογισμό. Αλλά αυτό δεν φαίνεται. Ποιο τμήμα οφείλεται σε μία επιλεξιμότητα των προγραμμάτων, τη δομή του ή σε δημοσιονομικά προβλήματα. Και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νέων κανόνων, όταν ε, τα τρία κοινοτικά θεσμικά όργανα διαπραγματεύτηκαν μεταξύ τους κανόνες, δεν ε, είχαμε μιλήσει καθόλου για την ε, εγκατάλειψη πρότασης της ανακοίνωσης. Τι γίνεται με αυτούς το επιπλέον τρίμηνο. Γιατί νομίζω ότι οι κοινοποιήσεις στους ενδιαφερομένους γίνονται πολύ πιο καθυστερημένα. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια επιχειρηματολογία γιατί άλλαξαν τα πράγματα εδώ. Και πιστεύω ότι θα πρέπει από κοινού να δείξουμε και με διαφάνεια ποιες θα είναι οι συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για το πρόγραμμα. Και είναι σημαντικό αυτό στις επικείμενες διαπραγματεύσεις του προπολογισμού με το Συμβούλιο. Κύριε Έλερ, εσείς ήταν ο εκπρόσωπος όλων των εισηγητών της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας, γι' αυτό και σας επέτρεψα να παραβείτε το χρόνο που δικαιούσατε. Αλλά οι υπόλοιποι λοιπόν, παρακαλώ να εμείνετε στο δίλεπτο που δικαιούστε. Η κυρία Καμπεσόν Ρουίς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσίαση που ήταν σύντομη, 12 λεπτά μόνο, αλλά εξαιρετικά διαφωτιστική. Εγώ έχω και δύο παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Μία τεχνική ερώτηση και μία πολιτική. Ποια είναι η γνώμη σας για την εφαρμογή του άρθρου 27 των κανόνων συμμετοχής για το άμεσο κόστος του προσωπικού που λαμβάνει επιδοτήσεις Κανονικά θα πρέπει να είναι εύκολ, οι προϋποθέσεις ε, για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ε, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 2020, ορίζοντας 2020, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μας λένε ότι το αντίθετο συμβαίνει και οι κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστούν τελείως ανεφάρμοστο το μέτρο αυτό, οπότε έχουν, πρόβλημα οι ερευνητές ό,τι αφορά τις ε, την αμοιβή τους και τις επιδοτήσεις. Μήπως ε, τι πρέπει να γίνει για να εφαρμόζεται η ερμηνεία των ε, αρχών σας ό,τι αφορά, των υπηρεσιών σας σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Επίσης, ε, για το τεχνικό έργο της Πρίμα δεν έχει οριμάσει αρκετά για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σύνδεσης για τη Μεσόγειο με βάση το άρθρο 185 της Συνθήκης. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά απρόθυμη. Και επικαλείται μάλιστα τρία επιχειρήματα. Λέει ότι είναι χρονοβόρη διαδικασία. Το γνωρίζουμε αυτό. Τέσσερις τουλάχιστον αποφάσεις στηρίζονται σε αυτό το άρθρο 185. Γι' αυτό και πέρασε 11 που είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Και η ανάληψη υποχρεώσεων αφορά περίπου 200 εκατομμύρια και συγχρηματοδότηση ένα τμήμα τους. Πιστεύετε ότι μία πρωτοβουλία κοινής, κοινού προγραμματισμού θα τα χρήσιμη εδώ. Γιατί σίγουρα οι ενδιαφερόμενοι έχουν εκδηλώσει την δέσμευσή τους και το ενδιαφέρον του και πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει οριμάσει για να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να εφαρμόσουμε και εμπράκτο το άρθρο 185 της Συνθήκης. Ευχαριστώ κύριε Χένκελ. <clears throat> Θα ήθελα να σχολιάσω ένα διαφορετικό ζήτημα. Ε, παραπονηθήκατε για τις περικοπές στον προϋπολογισμό. Εμένα με σοκάρει το ότι η θέση ε, του ανώτατου επιστημονικού συμβούλου καταργήθηκε. Δεν το καταλαβαίνω η Επιτροπή, ο Πρόεδρος δεν ενδιαφέρονται πλέον για την επιστημονική αλήθεια, τα επιστημονικά τεκμήρια. Βασιζόμαστε σε πολιτική ιδεολογία πλέον για να αποφασίσουμε ή θα εξακολουθήσουμε να βασιζόμαστε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, γιατί είναι και βασική ανησυχία και δική μου και της ομάδας μου, δεν ε, υπάρχει αυτή η θέση πλέον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για την επιστημονική αλήθεια ακόμη. Ναι ή όχι, το ελπίζω. Άλλα δύο ζητήματα. Αναφερθήκατε στο όργανο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τις πρώτες προσφορές ε, που λάβατε στην πρόσκληση υποβολής μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ε, οι μικρομεσαίες και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την ε, πρώτη κατανομή κονδυλίων. Δεύτερον, μιλήσατε για το πρόβλημα έλλειψης κονδυλίων Ταυτόχρονα η Eurostat στην έκθεσή της ξεκαθάρισε ότι περίπου το 2% του ΑΕΠ ε, διοχετεύεται στην έρευνα και την καινοτομία ε, από τα κράτη-μέλη και θα θέσω ένα ευρύτερο ερώτημα. Μήπως με τον ορίζοντα 2020 θα ασκηθεί και μία πίεση στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τους ευρύτερους στόχους που θέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πόσον και εφόσον ε, κάποια κράτη-μέλη δεν ξεπερνούν ε, το 3% για την έρευνα και την καινοτομία, να ρωτήσουν πώς θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε βάση το ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ κυρία Μπαρμπάρα Κουντρίτσκα. Ευχαριστώ. Ήθελα πρώτα απ' όλα Να σας συγχαρώ για το βραβείο που πήρατε. Είναι πολύ καλός ο τρόπος που συντάσσονται πλέον οι ενημερωτικές εκθέσεις. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου τώρα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Τι γίνεται με τη συμμετοχή, το μερίδιο τη της κάθε χώρας σε ό,τι αφορά το ορίζοντας 2020. σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη συμμετοχή των περιφερειών που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετά. Και ποιο ε, τμήμα των, ε, των, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ε, τη μερίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ε, τι ποσοστό είναι αυτό που για πρώτη φορά συμμετέχει στο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία για το μερίδιο των χωρών μελών και το ποσοστό των περιφερειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ορίζοντας 2020. Από τους πρώτους διαγωνισμούς μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι απλουστευμένες διαδικασίες και ευκολότερη πρόσβαση ε, επηρεάζουν ε, τους υποψηφίους και τους, τους παροτρύνουν να υποβάλουν πολύ περισσότερες προτάσεις. Ευχαριστώ κύριο Σιλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Διευθυντή για την εδώ παρουσία του ε, και τη σύντομη αλλά περιεκτική ομιλία του. Είναι κοινό αποδεχτών ότι το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την έρευνα και την κοινοτομία... που να δώσει όθηση στην οικονομία ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης σε μια περίοδο που είμαστε μέσω ε, ε, γενικότερης κρίσης. Ε, παράλληλα μπορεί να στηρίξει ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προωθήσει νέες θέσεις εργασίας αλλά κατά ένα μας να ενισχύσει την κοινωνική ανάπτυξη. Ήδη έχουμε κάποια προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι τις περικοπές που έχουμε στον προπολογισμό του 2015 σε έναν προπολογισμό που ήταν έτσι κι αλλιώ ε, κουτσουρωμένο κατά την άποψη του Κοινοβουλίου. Το δεύτερο έχει αποδειχτεί ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επειδή αναφερθήκατε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι ιδιαίτερα ε, πάρα πολύ δύσκολη λόγω των διαδικασιών. Ε, και το τρίτο σημείο είναι ότι ευνοούνται οι συνέργειε μεταξύ τη ακαδημαϊκής κοινότητα και του ιδιωτικού τομέα, όμω το πρόγραμμα μετατρέπεται πολλέ φορέ σε εργαλείο κατά την άποψή μα των μεγάλων πολυεθνικών, το οποίο βέβαια αναπτύσσεται βάσει των δικών του αναγκών και συμφερόντων αντί των αναγκών και των συμφερόντων τη κοινωνία. Τα ερωτήματα μου πολύ σύντομα. Τι μέτρα θα προωθήσετε για να ενισχύσετε περαιτέρω το πρόγραμμα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη κοινωνία. Το δεύτερο που δεν έχουμε μέχρι σήμερα απαντήσει είναι πώ θα απλοποιήσετε τι διαδικασίε χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδιαίτερα εκείνε που πλήττονται. Ήδη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την, ε, τον κορμό της οικονομίας της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ε, και το τρίτο, πώς αντιμετωπίσετε τις συνέπειες ε, που προκύπτουν λόγω της μείωσης των προπολογισμών. Ε, ποια μέτρα δηλαδή θα παρτούν ώστε να διατηρηθεί το πρόγραμμα ορίζοντας, ορίζοντας, ορίζοντας 2020 στο στόχο που έχει τεθεί από την αρχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Mr. Tamburano, would you like to say something? No, thank you. And Mr. Πρέπει να... Roger Helmer. Κύριος Ρότζερ Χέλμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον Γενικό Διευθυντή. Αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής ε, είναι ότι ε, Κακώς το Συμβούλιο περιορίζει τις δαπάνες και καλά κάνει το Κοινοβούλιο που ζητά επιπρόσθετα κονδύλια. ό συνήθως εδώ στο Κοινοβούλιο φαίνεται ότι και πάλι δεν έχουμε καμία επαφή με το ότι στην Ευρώπη ε, όλοι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότατη ανεργία, δημοσιονομικές ε, περικοπές, ε, ε, την χρηματοοικονομική κρίση. Πώς λοιπόν περιμένετε εσείς ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθήκων να συνεχίσουμε να δαπανούμε τέτοια κονδύλια. Σίγουρα η δουλειά μας δεν είναι όταν προσπαθούν όλοι να ελέγξουν τις δαπάνες να ζητούμε επιπρόσθετα κονδύλια. Η δουλειά μας είναι να ε, δαπανίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα κονδύλια που παραμένουν διαθέσιμα και από το αντί να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια και να τα αφήνουμε να χάνονται μέσα από τον γραφειοκρατικό έλεγχο των Βρυξελών, καλό θα ήταν και αποτελεσματικό και με πιο κοντινό με την πραγματικότητα θα ήταν να αφήναμε αυτά τα κονδύλια να τα διαχειρίζονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε εθνικό ή ακόμη καλύτερα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και όχι εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ να σας ζητήσω να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων ε, σε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ο κύριος Σμίτς. Ας αρχίσω από το τελευταίο ζήτημα. Μετά από ε, μακρύς διαπραγματεύσεις καταλήξαμε σε συμφωνία για τον ορίζοντα 2020 ε, στα 80 δις συγκεκριμένα. Αυτή ήταν η συμφωνία του ε, Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και όταν μετά από μια δημοκρατική διαδικασία καταλήγουμε ε, σε ένα σημαντικό όργανο που βασίζει στις αρχές της ευρωπαϊκής προστάμενης αξίας και της οπικουρικότητας ε, και προκύπτει ένα ποσό 80 δις, ε, σημαίνει ότι έχουμε τα χρήματα για να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό. Δεν ζητάμε πρόσθετα κονδύλια. Αυτό που ζητάμε είναι Αυτά τα κονδύλια να τα λάβουμε ε, και είναι τα κονδύλια επί των οποίων συμφώνησε το Κοινοβούλιο μετά από πάρα πολύ μακρές διαπραγματεύσεις. Ε, και ξέρετε η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία έχει αποδειχθεί από διάφορα ε, προγράμματα όπως το ίτερ παραδείγματος χάρη και η χώρα σας ξέρετε είναι μία, ένας από, μία από τις ε, σημαντικότερες χώρες δικαιούχους του 7ου προγράμματος πλαισίου και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερο αποδέκτης των κονδυλίων που διατίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έρευνα και για την καινοτομία. Α ε, προχωρήσω στι υπόλοιπε παρατηρήσει. Κύριε Έλλερ, χαίρομαι πολύ που θα υπάρχει μόνιμη επιτροπή ε, για τον ορίζοντα 2020. Φυσικά, με μεγάλη χαρά θα σα δώσουμε ό,τι χρειάζεστε. Στοιχεία, στατιστικά, προγνωστικά, εκτιμήσει, οτιδήποτε να μα ζητάτε. Ε, μιλήσατε για την υπερκάλυψη, το θέμα της ε, υπερκάλυψης ε, στην υποβολή, πρόσκληση υποβολής προσφορών. Πώ Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Πρώτον, είναι ε, δημοφιλέστατο το πρόγραμμα και είναι, εξαιρετικά δημοφιλές στην επιστημονική κοινότητα. Δεύτερον, χάρη στην απλούστευση, ακόμη και για νοησερχόμενους, δεν έχουμε τόσους πολλούς φραγμούς και είναι πάρα πολύ ευκολότερη η πρόσβαση. Και τρίτον, Έρχονται πολλοί, αυτό με ε, δυσαρεστεί, διότι έχουν κοπεί, περικοπεί τα εθνικά κονδύλια. 600 ε, εκατομμύρια ε, περιέκοψε η Ισπανία από τον ε, προϋπολογισμό της για την έρευνα και έρχονται στις Βρυξέλλες οι ερευνητές. Ε, Βεβαίω αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να βασιστούν σε ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, σε ευρωπαϊκή συνεργασία. να ασχολούμαστε με εθνικά προγράμματα. Τι κάνουμε τώρα για να καλύψουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της υπερκάλυψης. Ε, υιοθετούμε ε, την διαδικασία σε δύο χρόνους. Ε, σε μία πρώτη φάση υποβάλλονται οι προσφορές και όταν κριθεί η κατάλληλη η προσφορά περνάει στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή από το, το 20% θα περάσει στο δεύτερο στάδιο και από όλες τις προσφορές και στη συνέχεια το 30% θα λάβει επιδότηση. Το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο είναι ένας άλλος ενδιαφέρον μηχανισμός. Αν υποβάλλεται μία προσφορά, ε, μάλλον χαμηλής ποιότητας ε, και αυτό αξιολογηθεί έτσι από το Συμβούλιο Ομοτήμων, πρέπει να περιμένετε δύο-τρία χρόνια πρωτού υποβάλλετε και πάλι προσφορές. Ε, και επειδή είναι τόσο δημοφιλέ το πρόγραμμα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της υπερκάλυψης. Ε, στις πρώτες ε, συμβάσεις μπορέσαμε να τηρήσουμε το οχτάμινο που ζήταγε το Κοινοβούλιο και νομίζω για του δικαιούχους και για μας είναι σημαντικό να υπάρχει πολύ καλή ενημέρωση γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος και θα πρέπει όλοι να ενημερωθούν. Κυρία Κάπρισον, μας ε, ε, Μιλήσατε για τους συντελεστές χρηματοδότηση. Στον ορίζοντα 2020 ε, προκρίναμε για όλους τους συμμετέχοντες ενιαίο συντελεστή για χάρη της απλούστευσης. 20% 25% του έμεσου κόστους ε, καλύπτουμε ε, και ε, για την έρευνα και 70% για τα υπόλοιπα για τα πάγια, για, τα, για τις ουσιαστικές δαπάνες και 20% για τα πάγια. Θα καλύπτονται πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αυτοί που ενδεχομένως θα έχουν πρόβλημα θα είναι αυτοί που έχουν υποδομές μεγάλης κλίμακας και ε, όντως θα βρούμε μια ρύθμιση, ένα μέρος του έμεσου κόστους να ε, μεταγραφεί στην κατηγορία άμεσου κόστους. Ε, εν γέννη πάντως οι διατάξεις είναι ικανοποιητικέ για τους συμμετέχοντες. Ε, κύριε Χένκερ, μας μιλήσατε για τον Ανώτατο Επιστημονικό Σύμβουλο και την θέση αυτή και μιλήσατε για τον πρόεδρο. Φυσικά, ο πρόεδρο είναι απόφαση για την πλήρωση αυτή τη ε, χειρεύουσα θέση, χειρεύουσα διότι δεν έχει καταργηθεί. μετά το πέρασε της θητείας ε, της δεύτερης επιτροπής Μπαρόσο παραμένει κενή ε, διότι μεταρρυθμίζονται οι διοικητικές δομές. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για κατάργηση της θέσης ακόμη. Έχει λήξει η θητεία προς το παρόν και ε, μετά τις προϋποθέσεις διαπραγματεύσεις θα δούμε πώς θα καλυφθεί η θέση. Είμαστε πεπισμένοι πάντως πώς βασιζόμαστε ε, σε επιστημονικά στοιχεία, αντικειμενικά αποστημονικά στοιχεία και όχι σε υποκειμονικές εκτιμήσεις. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ε, η επιστημονική τεκμηρίωση θα παραμείνει βάση των αποφάσεων μας. Ε, ο κύριος Δεμπέκερ αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να ε, διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων. Τι κάνουμε για αυτές λοιπόν. Πρώτα απ' όλα 20% του προϋπολογισμού είναι για τις μικρομεσαίες. Δεύτερον έχουμε ε, ειδικό όργανο για τις μικρομεσαίες ε, με πολύ καλό σημείο εθνικών σημείων επαφής. Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις και τρίτον απλούστευση. Τα μέτρα απλούστευσης διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων. Κυρία Κουντρίτσκα, σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Όπως όλοι, ε, ανησυχείτε κι εσείς για την αριστεία σε εθνικό επίπεδο και εσείς η ίδια αναλάβατε την πρωτοβουλία του Teaming Action των ομάδων στα πλαίσια του ΡΙΤΟ 2020 Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χάρη στην απλούστευση, ε, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, θα έλεγα ότι με το που συσταθεί η δική σας μόνιμη Επιτροπή θα δίνουμε στατιστικά στοιχεία, θα σας διοχετεύουμε στατιστικά στοιχεία για να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα ε, της κατάστασης ε, και... Μία άλλη σημαντική ερώτηση ήταν τα έξοδα, τα, οι δαπάνε 2% για την ε, έρευνα και την καινοτομία. Πολλοί μιλάνε για αυτά τα ζητήματα, αλλά λίγοι επενδύουν. Τώρα είμαστε στο 2% του ΑΕΠ και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό το ρίζο το 2020 για την χρηματοδότηση από πλευρά των κρατών. δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να υπομισθούν τα κράτη-μέλη την ευθύνη του και να επενδύσουν στο μέλλον. Αυτό που με τρομάζει είναι ότι οι δαπάνε ε, τη Κίνα ε, αυξάνονται κατά 22% το χρόνο. Η Κορέα ε, ε, ξοδεύει το 5% του ΑΕΠ ε, στην έρευνα και στην καινοτομία. Θα πρέπει να λειτουργήσει ως κλίση αφύπνισης, να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε και όχι μόνο να μιλάμε για την έρευνα και την καινοτομία. Ευχαριστούμε. 10-11 έχω στο κατάλογο των ομιλητών. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα κλείσει τώρα ο κατάλογος των ομιλητών. Έκλεισε μάλλον. Και... Ένα λεπτό. Εκαστός, γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε μέχρι τις 5. Γκρίφιν, ένα λεπτό. Ε, thank you. Σας ευχαριστώ πρόεδρε ως αντιπροσωπή του Ηνωμένου Βασιλείου και εμείς ε, ανησυχούμε σχετικά με το κόστος ε, της, ε, των επιστημονικών συμβούλων. Ε, χαιρόμαστε όμως που μιλήσατε για την αριστεία. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι και αυτοί που αποκλείονται από την αγορά εργασίας να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υψηλά αμοιβόμενες θέσεις στο μέλλον. Τώρα, ε, πώς θα γίνει διαφοροποίηση ανάμεσα στο Horizon 2020, τα διαρθρωτικά ταμεία, ε, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση, πώς μπορούν και να συνδυαστούν όλα αυτά, τι είδου ε, μέτρα πρέπει να λάβουμε για να μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο. Πολύ ωραία, ο κύριος Γκεμπράντη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κύριε Σμίθ που ήρθατε και φίξατε και τα θέματα του προϋπολογισμού γιατί ανησυχούμε ιδιαίτερα ακούγοντας ότι θα έχουμε, αν συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, ε, δηλαδή δεχόμενη τις συμβουλές του Συμβουλίου ένα κενό της τάξης του 40%. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Συνήθως μιλάμε για θέματα προϋπολογισμού ε, κάτω από το πρίσμα της μακροοικονομίας. Είπαμε το πρόβλημα του 2014, το λύσαμε μετακυλίοντας κάποιες προτάσεις για την επόμενη χρονιά όμως οποτεδήποτε μιλάω σε εταιρείε, σε φορείς, όλοι αυτοί μιλάνε για μια αξιόπιστη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες δαπάνες ε, που δεν πληρώνονται και αναβάλλονται. Μήπως μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος τι θα συμβεί ακριβώς αν τελικά το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τις ε, πληρωμές που είναι απολύτως απαραίτητες. Εγώ έχω μια ερώτηση για θέματα υγείας σε σχέση με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Κατά την προηγούμενη θητεία δεν αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία ε, σε ένα μεγάλο πρόβλημα, την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Αύριο είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για αντιβιωτικά. Αν λοιπόν δεν κάνουμε έρευνες και δεν βρούμε νέους τρόπους για να αντιμετωπίζουμε τα αντιβιωτικά ε, και αν δεν κάνουμε και έρευνα για νέα αντιβιωτικά, τότε θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στον τομέα της φροντίδας για λόγους υγείας. Και αυτά ε, συνδέονται άμεσα και με θέματα παραγωγής γιατί αλλάζουν και οι ε, χρειαζόμαστε άλλα αντιβιωτικά για να του αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν ίσως ε, πρέπει κατά επόμενα πέντε έτη ε, να προβληθεί περισσότερο το θέμα αυτό, διότι δυστυχώς φοβάμαι κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν και δεν θα μπορέσουμε να τους θεραπεύσουμε στα κέντρα υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που είναι εν μέρει αισιόδοξες και εν μέρει απεσιόδοξες. Φυσικά απεσιοδοξία από τον προπολογισμό, αισιοδοξία από την ε, απλοποίηση που προχωρεί. Η τραγική πάντως ε, πλευρά αφορά το πώς θα διαχειριστούμε τις ελλείψεις ε, κονδυλίων. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας ιδιαλλαγής και έχουμε προβλήματα όχι με το 2015 αλλά και για απλήρωτους λογαριασμούς το 2014. Οπότε είναι εύλογες οι ανησυχίε των δικαιούχων, ε, ιδιαίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φαντάζομαι θα πρέπει να απασχολεί, απασχολήσει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η έλλειψη χρημάτων ε, και να διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν. Γιατί δεν θα έχουμε μόνο το χρόνο πρόβλημα και φέτο. Ο κύριο Ζωρίνιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά και να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή να εξάρω τη σημασία που έχει η στενή συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προκειμένου να καταδείξουμε την, ε, το παράλογο των ε, περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό. Αυτή η σχιζοφρένεια στη ρητορική που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και μάλιστα ήδη από το Δεκέμβριο έχει προαναγγελθεί και ένα επενδυτικό πρόγραμμα για ορισμένου τομείς που είναι και προτεραιότητες του Ορίζοντα 2020. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία μεταξύ έργων και λόγων και διαφορά. Για πολλά χρόνια συνεργαστήκαμε με ερευνητικά κέντρα, με ομίλου και διαπιστώσαμε ότι υποβλήθηκαν πολλέ εξαιρετικέ προτάσει και έχουμε πολλού πόλου αριστείας. Καλή αυτή η πόλη αριστείας, αλλά δεν μα φέρνουν σε πρωταγωνιστική θέση στο διεθνή στίβο. Και όταν έχουμε κανόνες πολύ πιο φιλικές προς τις ε, επιχειρήσεις δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε και φιλικούς κανόνες προς την καινοτομία. Αλλιώς θα μείνουμε πίσω σε σχέση με τους ε, άλλους εταίρους μας. Η κυρία Βέρνερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά, έχω μια καθαρά πρακτική φύση ερώτηση. Δηλαδή, στο πλαίσιο του εργαλείου για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι εταιρείε των οποίων απορρίφθηκαν αιτήσει δεν παίρνουν ε, έκθεση αιτιολόγηση και αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λόγω του ότι υπάρχει αυτό το πολύ μικρό ποσοστό επιτυχία που αναφέρεται σε σχέση με τι αιτήσει, προφανώ οι επιχειρήσει που απορρίπτουν οι αιτήσει του αισθάνονται απογοητευμένε και δεν κάνουν δεύτερη προσπάθεια. Ε, γιατί δεν ενημερώνονται το γιατί όπως σας είπα απορρίφθηκε η αίτησή τους και γιατί δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές. Η Κομισιόν λοιπόν γνωρίζει αυτά τα προβλήματα και αν ναι τι προτίθεται να κάνει. Ευχαριστώ κύριε Σάντερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή. Έχω μία παρατήρηση ε, πιστεύω, όπως και προλαλήσαντες, ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε την ε, διαδικασία της απλούστευσης. Γιατί, γιατί όπως σας λένε και οι ερευνητές, ε, πολύ περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να σχεδιάσουν το πρόγραμμα και να το δρομολογήσουν καθημερινά από ότι χρόνο αφιερώνουν στην ίδια την έρευνα. Επίσης είναι τεράστιο το δημοσιονομικό κόστος των ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων γιατί οι ερευνητές αναλαμβάνουν και το διοικητικό φόρτο γιατί δεν έχουν άλλον για, να το, για να το αναθέσουν αυτό το διοικητικό φόρτο. Γι' αυτό νομίζω ότι επήγει η διοικητική απλούστευση. Ο κύριος Τσούλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος 2020 μιλήσαμε πάρα πολύ για την αποκαλούμενη στρατηγική εξειδίκευση ε, έτσι ώστε οι τοπικές ε, αρχές ε, να μπορούν να χρηματοδοτούν τους τομείς εκείνους που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα λοιπόν που κάνω είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιο τρόπο στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς για να χρησιμοποιούν καλύτερα τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων έτσι ώστε να παρουσιάζουν περιπτώσεις αριστείας και να μπορούν με τον τρόπο αυτό να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα κονδύλια του προγράμματος ορίζοντας 2020. Ο εισηγητής μας, πολύ σύντομα παρακαλώ. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε λιγάκι πολύ συγκεκριμένα τους αριθμούς. Τι ακριβώς σημαίνουν οι περικοπές ε, του προπολογισμού για το ορίζοντας 2020. Καλό αυτό που επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά είναι και επικίνδυνο. Λείπουν 6 δις, ε, έλειπαν και άλλο ένα 1,1 δις. Ε, γι' αυτό λοιπόν, εάν από τα 14 έχουν ήδη δοθεί τον 9,3 καταλαβαίνετε μέχρι το 2007 ε, θα είμαστε πολύ πιο κάτω κάτω από τα 6 που χρειαζόμαστε αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα χρειαζόμαστε ως ένα επιχείρημα που μπορούμε, να μπορούμε να προβάλλουμε στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο Ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι για τις ερωτήσεις Συνέργειες μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και ορίζοντα 2020 το επισήμαναν πολλοί ομιλητές και χαιρόμαστε γιατί ε, στα διαρθρωτικά ταμεία όχι μόνο έχουμε κονδύλια για υποδομές μεταφορών, αλλά και για τη γνώση, για ε, εκολαπτήρια έρευνας, για συνεργασία με τα πανεπιστήμια, για να δημιουργήσουμε πραγματικά τη σκάλα προς την αριστεία, για να μπορέσουμε να ανέλθουμε την αριστεία. Νομίζω ότι από αυτήν την άποψη έχουμε καλή συνέργεια και έχουμε καλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, Ισπανία και Ιρλανδία χρησιμοποίησαν και οι δύο τα διαρθρωτικά ταμεία για να γίνουν ε, χώρες της γνώσης, γιατί επένδυσαν όχι μόνο σε υποδομές μεταφορών, σε αυτοκινητοδρόμους και σε αεροδρόμια, αλλά για την εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων τους και τον ερευνητικό τους κέντρο. Μερικοί με ρώτησαν ποιε είναι οι συγκεκριμένε συνέπειε των δημοσιονομικών περικοπών. Ε, αναφέρθηκαν από τον αρμόδιο, από τον αρμόδιο επίτροπο πόσες, ε, πόσες κονδύλια μας λείπουν από το πρόγραμμα Ρικιουρί, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις θερούνται χρηματοδότησης. Είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία. Ο κύριος Γκεμπράντη με ρώτησε αυτό στην πράξη τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν εγκρίνουμε ένα σχέδιο με συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα και δεν μπορούμε να το προχρηματοδοτήσουμε, δεν θα μπορέσουν οι αρμόδιοι του προγράμματος ε, να προσλάβουν προσωπικό, να ξεκινήσουν το πρόγραμμα. Αυτές είναι οι έμπρακτες συνέπειες. Πολύ ζωφερές λοιπόν, ιδιαίτερα σε ένα σημαντικό κλάδο όπως είναι η επιστήμη και η καινοτομία. Αύριο είναι η μέρα των αντιβιωτικών, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την ε, μικροβιακή ε, αντοχή στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό με την φαρμακευτική βιομηχανία και τα ερευνητικά κέντρα, ε, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε 300 εκατομμύρια για να διερευνήσουμε εναλλακτικέ λύσει. Γιατί αυτό το πρόβλημα τη μικροβιακή ε, αντοχή στα αντιβιωτικά επηρεάζει άμεσα του πολίτε. Και αύριο θα σα δώσουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση υπόδειγμα για τέτοιου είδου ε, προγράμματα. Επίσης, είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί κάθε χρόνο εξαντλούμε τα κονδύλια μας και πέρυσι, κύριε Λεβαντόφσκι, όσο ήσταν αρμόδιος για τον προϋπολογισμό ε, επίτροπος, ε, είπατε ότι το πρόγραμμά μας είναι παράδειγμα προς για απόλυτη εκταμείευση των κονδυλίων. Γιατί πέρυσι ε, μας έμειναν 280, 280 σε ένα πρόγραμμα εκατομμύρια, Εμεί μέχρι το τελευταίο ευρώ εκταμιεύουμε τα κονδύλια που έχουμε διαθέσιμα και νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το feedback που δίνουμε στους ε, υποβάλλοντες αίτηση. Ακριβώς επειδή κατακλυζόμαστε από προτάσεις, δεν προλαβαίνουμε να στείλουμε ε, εκτενείς επιχειρηματολογίες για την απόρριψη. Προσπαθούμε όμως να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή και στην επόμενη διαγωνισμό να στέλνουμε πιο λεπτομεριακό σχολιασμό μία απόρριψη. Γιατί όσοι έχουν υποβάλει, όσοι έχουν μπει στον κόπο να υποβάλουν προγράμματα, νομίζω ότι δικαιούνται και αξίζουν να εξηγήσω σε περίπτωση που δεν επιλέγουν αυτά. Αυτά και ελπίζω να μην παρέλειψε καμία πρόταση. Όπως είπαμε επανειλημμένος, νομίζω ότι το όταν χρησιμοποιούμε κονδύλια στον, στον ορίζοντα 2020 δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο δαπανούμε κονδύλια, αλλά επενδύουμε για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, για τα πιο φλέγοντα ζητήματα για του συμπατριώτες μα. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα στι 7 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει η έκτη διάσκεψη κορυφής για τη γνώση και την καινοτομία. Παρουσία τριών επιτρόπων. Ε, για την ε, έρευνα και καινοτομία, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωργία. Θα έχουμε την παρουσία τριών ολοκένουργων επιτρόπων μας και θα συζητήσουμε για την καινοτομία και για το πώς ε, θα δαπανίσουμε καλύτερα τα κονδύλια μας ώστε να πιάσουν τόπο σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσία σας και για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Θα έχουμε τακτικές επαφές ε, την υπόλοιπη, υπόλοιπη πενταετία, γιατί πραγματικά για το μέλλον χρειαζόμαστε τέτοιες τακτικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. So, nothing. Okay. Perfectly We are Τέλεια οργάνωση. Τέσσερις ακριβώς και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Τις ψηφοφορίες για την ακριβή, γιατί έχουμε δύο ψηφοφορίες. Η πρώτη αφορά την ανανέωση της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ουκρανίας. Πολύ σημαντικό θέμα, γιατί η παλιά συμφωνία εξέπνευσε στις 7 Σεπτεμβρίου. Στις ε, 7 συγγνώμη Νοεμβρίου του 2014, πριν από ένα δεκαήμερο δηλαδή. Ε, ολοκληρώθηκε η, η συμφωνία που αφορά εντατικοποίηση, συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας ε, προς ε, όφελος επιστημονικής κοινότητας αλλά και των πολιτών. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτα θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργούν οι συσκευές. Μια δοκιμαστική λοιπόν ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργούν οι συσκευές. Δεν προβλέπεται μυστική ψηφοφορία έτσι. Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία, πολύ σημαντική. Θα σας δώσω μία ερώτηση. Για παράδειγμα, σας αρέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, απαντήστε, ψηφίστε. The vote is open. Okay, we will see. Uh, the vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απλή ερώτηση. Αχ, συνάδελφοι, η η ερώτηση ήταν σαφής, αλλά η απάντηση δεν είναι και πολύ σαφής. Θα, θα προτιμούσα κάπως διαφορετικά συμπεράσματα. Πάντως, αμέριστη υποστήριξη προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωραία, τα μηχανήματα λειτουργούν. Τώρα ψηφίζουμε κανονικά ανανέωση συμφωνία επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ουκρανία. Ψηφοφορία ηλεκτρονική, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, Προμπάτο που λένε και οι Ιταλοί. Δεν τα είπα τέλεια και η προφορά μου. Δεύτερο θέμα, συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικού σκοπού μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των κρατών μελών τη αφενό και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αυτό απρομπάτω. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Η οργάνωσή μας είναι εντυπωσιακή. Δεύτερη φορά που το διαπιστώνουμε σήμερα. Περάμε στο σημείο 6. Δημιουργία και λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση κάποιες οδηγίας. Η μας είναι ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ κύριε Ταγιάννη, έχετε ένα πεντάλεπτο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω τη θέση μου ότι είμαι υπέρ αυτών των μέτρων. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει μια ισχυρή Ευρώπη που να μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Και αυτό το σύστημα ε, της ε, ανταλλαγής εκπομπών. Αυτό είναι ένα σύστημα αποτελεσματικό. Έχουμε το 40% των θερμοκηπίων αερίου το, μέχρι το 2030 που θα πρέπει να μειωθεί κατά 40%. Πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει και έναν άλλο στόχο που όμως ε, το Συμβούλιο επίσης τον υιοθέτησε βέβαια και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή το 20% του καθάριστου εθνικού προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το 2020 θα πρέπει να προέρχεται από την βιομηχανία. Έτσι λοιπόν πρόκειται σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό τον ε, τομέα για ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό για το βιομηχανικό μας σύστημα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια ισορροπία και παράλληλα βέβαια να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και την κλιματική αλλαγή αλλά και την επανεκβιομηχάνηση την αναγέννηση της βιομηχανίας. Βεβαίως και πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το γάμο ανάμεσα στη βιομηχανία και τις ε, ε, πολιτικές για το κλίμα. Όμως αυτός ο γάμος δεν πρέπει να είναι εις βάρος της βιομηχανίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι ο βασικός μας στόχος που είναι να ξεπεράσουμε την κρίση, άρα δηλαδή πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Είναι επίση αλήθεια ότι υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός και αυτό ότι αυτό είναι η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα πριν από κάποιες μέρες ε, στον αγώνα κατά της ε, κλιματικής αλλαγής. Βέβαια αυτός είναι ένας μακρόπνο στόχος και καθότι λείπει μια οικουμενική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, επειδή λείπει λοιπόν αυτό, είναι δύσκολο για μας να προχωρήσουμε. Ως εκ τούτου οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά ε, την προστασία των δικών μας υποθέσεων. Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε μειώσει βέβαια τις εκπομπές μας, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 18%, ήταν το 14% το 2010 και σήμερα είναι μόνο το 10% των ε, παγκόσμιων εκπομπών. Και ε, υποτίθεται ότι ε, το 2050 θα έχουν μειωθεί περαιτέρω περίπου στο 8%. Πρέπει βέβαια να υπάρχει ένα αποθεματικό σταθεροποιητικό για την αγορά. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, κυρίως μετά το περίφημο black loading. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε αυτό το σύστημα να ε, βοηθήσει κυρίως ε, τις χώρες ε, που αγωνίζονται πραγματικά για την κλιματική αλλαγή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ε, να λαμβάνεται υπόψη, να λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές του διοξιδίου, αλλά υπάρχουν πολλές δυσάρες εκπλήσεις, όπως μια αυστριακή, η Vestalpin, μια εταιρεία, αποφάσισε να μεταβεί στις ΗΠΑ και βεβαίως είμαι αναγκασμένος και να επενθυμίσω και την πολύ δυσάρεστη ε, περίπτωση δική μου της χώρας την παραγωγή ε, από την Σικελία που και αυτή η βιομηχανία έκλεισε. Εκείνο λοιπόν που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε είναι τα κοσμήματά μας, τα βιομηχανικά μας κοσμήματα να φεύγουν και φεύγοντας χάνονται βέβαια και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Θεωρώ, θεωρώ ότι το σύστημα θα πρέπει να προσαρμοστεί κυρίως με βάση κάποια ε, συγκεκριμένα κριτήρια. Τον Ιανουάριο, ε, στο πλαίσιο του, ε, του 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε την υπάρχουσα στάθμι των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα και κατόπιν μετατέθηκε μέχρι το 2019. Ε, τους τελευταίους μήνες βεβαίως είδαμε ότι λαμβάνονται και συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο την ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανεκβιομηχάνηση αλλά και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Μαρτίου και Οκτωβρίου που επανεπιβεβαιώνουν την επανεκβιομηχάνηση ως το κέντρο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με στόχο κυρίως να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μεταποιητικός τομέας. Εκείνο που θέλω να σας επισημάνω και που θα το συζητήσουμε σήμερα αλλά εντάξει θα μπορέσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις τις επαναλάβουμε και κατά τις επόμενες μέρες. Ε, έλεγα λοιπόν ότι η δική μου η πρόταση είναι προς αυτή την κατεύθυνση και υπογραμμίζει κυρίως το θέμα της ανταγωνιστικότητας γιατί είναι καθοριστική σημασίας. Τη δική μου την εισήγηση που σας την έχω καταθέσει την επικεντρώνω σε πέντε σημεία. Το πρώτο αφορά τις ε, βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν περαιτέρω. Και αυτό το εργαλείο δυστυχώς ε, επιβεβαιώνει ή αυξάνει την ανασφάλεια. Για να το αποφύγει κανείς αυτό θα πρέπει να υπάρχουν 100% δωρεάν ποσοστώσεις μέχρι το 2030. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορεί να προσαρμόζεται με το επίπεδο παραγωγής που υπάρχει και όχι κάποια συγκεκριμένα κριτήρια καθορισμένα εκ των προτέρων όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά το κόστος ενέργειας που επιβαρύνει μέχρι και 40% το κόστος της παραγωγής στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Στην Ευρώπη είναι από τα υψηλότερα που υπάρχουν στον κόσμο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη επιθυμεί να μειώσει κατά 38% το κόστος ε, της ε, ενέργειας, ενώ ε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπήρξε μεγαλύτερη μείωση λόγω του σχιστολιτικού αερίου. Θεωρώ λοιπόν ότι αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις χώρες παραγωγούς που δυστυχώς όμως βέβαια δεν σέβονται αυτό τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής πρέπει να βρούμε έναν ισόρροπο οργανισμό για να υπολογίζουμε και το έμεσο κόστος και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας κατά νου ότι υπάρχουν και κάποια τεχνολογικά όρια ε, και το είναι δύσκολο να υπάρξει μια οικουμενική συμφωνία, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε πάντα κατά νου ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε, πρέπει να παρεμποδίσουμε τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να δώσουμε κίνητρα για την καινοτομία που θα οδηγήσουν στο να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και καθαρές ε, τεχνολογίες. Εγώ προτείνω αυτά που εισπράττουμε από το σύστημα της ανταλλαγής εκπομπών να τα επανεπενδύσουμε στην ανάπτυξη και την τεχνολογία. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Πολύ σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκρίφιν τώρα από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για την ε, ε, θέση που μας παρουσίασε σε σχέση με το μηχανισμό σταθεροποίησης των αγορών για το σύστημα εμπορίας ε, ρήπων ε, βάσει της πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε όλοι, δεν καταφέρνει το τωρινό σύστημα ETS να υπερπηδήσει το πρόβλημα της υπερβολικής προσφοράς αδειών. Τάχιστα, επιγόντως, πρέπει να αναλάβουμε μια δράση, ώστε ο μηχανισμός να μπορέσει να ελέγξει τις εκπομπές και να οδηγήσει σε επενδύσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο μηχανισμός σταθεροποίησης αγοράς μπορεί να αποδειχθεί το σωστό εργαλείο μόνο όμως εάν δώσουμε σωστό προσανατολισμό αλλά και πεδίο εφαρμογής. Πρώτον, η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί. Το ταχύτερο που θα αρχίσει, το, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι για να ε, καλύψει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της υπερβολικής προσφοράς αδειών. Εάν έχουμε το σωστό όργανο στα χέρια μας, γιατί να περιμένουμε και να μην το εφαρμόσουμε αμέσως. Το 2017 ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα ήταν η καταλληλότερη ημερομηνία έναρξης. Ε, δεύτερον, θα πρέπει να καταργηθούν οι άδειες που έχουν προσωρινά αποσυρθεί από την αγορά με το backloading. Εάν ε, προσπαθούμε να καλύψουμε ευρύτερα το ζήτημα της ε, υπερπροσφοράς, ε, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε και στη συνέχεια να επανεισάγουμε αποσυρθεί, αποσυρθήσεις άδειες στην αγορά. Βάσει τη πρότασή ε, του εισηγητή πιστεύω ότι είναι ε, καλύτερο να ξεκαθαρίσουμε τον στόχο του κανονισμού και να προσδιορίσουμε το πλαίσιο. Οι τροπολογίε ε, που έχουν κατατεθεί προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω δεν είναι πρόσφορες. Μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014 για το συνολικό τρόπο ευρωπαϊκό πλαίσιο του 2030 θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ονομοθεσία να επηρεάσει θετικά το μέλλον μας. Ας χρησιμοποιήσουμε τον κοινό νου. Ας δράσουμε τάχιστα και ας δράσουμε αποτελεσματικά με ξεκάθαρους στόχους. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Μέρος του ECR ο κύριος Τοσενόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ αντικαθιστώ τον κύριο Γκρομπάρτσικ από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικού που δυστυχώς κολλείεται και μου ανέθεσε να παρουσιάσω εγώ τις απόψεις του. Ο κύριος Γκρομπάρτσικ λοιπόν είναι ευγνώμων προς τον κύριο Ταγιάννη για την προσέγγιση του και κυρίως γιατί επισημαίνει κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονό δηλαδή ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκή ένωση στο σύνολό τη. Γιατί αν η διαδικασία του backloading, της μεταφοράς δικαιωμάτων δημιουργικής εκπομπών σε μεταγενέστερο χρόνο ε, εφαρμοστεί με ακραίο τρόπο, θα οξύνει τα προβλήματα στη βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μία συζήτηση που κάναμε πριν από ένα περίπου χρόνο στην Επιτροπή μας. Ήταν πραγματικά μία σφοδρή συζήτηση, πολύ φορτισμένη, για το σύστημα αυτό. Και ήταν και μία προειδοποίηση για το όλο σύστημα εμπορίας εκπομπών και το θέμα της αδειοδότησης. Συμφωνώ με τον κύριο Ταγιάννη ότι η διαδικασία του backloading είναι σημαντική, σημαντικό, σημαντική για την βιομηχανία που χρειάζεται ένα προβλέψιμο σύστημα. Θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε την αγορά για να αποφύγουμε την τη δημιουργία συμπληρωματικού κόστους για τη βιομηχανία. Έχουμε ήδη πρόβλημα υψηλών ενεργειακών τιμών που ούτως ή άλλως κάνει τη ζωή δύσκολη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να απλουστεύσουμε τα πράγματα και να βοηθήσουμε τη βιομηχανία. Και επίσης να προωθήσουμε την πρόοδο με ορθολογικό τρόπο. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή του συστήματος, να ενημερωνόμαστε στην Επιτροπή, γιατί ξέρω ότι γίνονται προσωμιώσεις, ε, συντάσσονται πίνακες. Το παρελθόν όμως οι προσωμιώσεις που έγιναν ε, δεν μας έδωσαν σωστές προβλέψεις για το μέλλον. Να αποφύγουμε τέτοια σφάλματα στο μέλλον, παρακαλώ. Είχαμε παρόμοια προβλήματα και στο παρελθόν, γιατί αν δεν είχαμε προβλήματα στο παρελθόν δεν χρειαζόταν να γίνει η σημερινή συζήτηση. Πάντω, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή μα, τον κύριο Ταγιάννη, γιατί πραγματικά υιοθέτησε μια πολύ λογική και συνετή προσέγγιση. Ο κύριος Φέντερλεκ, εκ των φιλελευθέρων. Θα είμαι Σουηδός, δηλαδή θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα μπω στο ψαχνό απευθείας. Έχουμε ε, διάφορες ανησυχίες με το κείμενο του κυρίου Ταγιάννη που τώρα συζητείτε και θα διαπιστώσετε ότι διαφοροποιούμε τη θέση μας. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε δεν θα θέλαμε το έγγραφο της ΙΤΡΑ να επικεντρωθεί μόνο στο σταθεροποιητικό αυτό μηχανισμό. Ο κύριος Σταγιάννη ε, μιλάει μέσα στο κείμενο και για την ε, διαρροή άθρακα. Ε, όντως θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγέ, αλλά να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα όταν θα γίνει η αναθεώρηση του συστήματος και ας αφήσουμε μόνο τον ε, σταθεροποιητικό αυτό μηχανισμό στο έγγραφο. Δεύτερον, όπως και οι σοσιαλιστές ε, θέλουμε το 2017, ε, το αργότερο 2018 για πρακτικούς λόγους να αρχίσει να ισχύει το σύστημα, οι χαμηλές τιμές στην αγορά είναι μια ε, αυταπάτη ε, για τις επιχειρήσεις ε, διότι τους δίνουν μια πλημελή εικόνα για τις τιμές σε σχέση με το 2021 και αν συνεχίσει το σύστημα όπως έχει τώρα θα πληγούν πολύ σοβαρότερα οι επιχειρήσεις, δεν θα μπορούν να προσαρμοστούν στις διαφοροποιημένες τιμές ε, το 2021 και γι' αυτό θα θέλαμε ε, νωρίτερα να αρχίσει να ισχύει το σύστημα 2017, άντε 18, ε, όπως και οι σοσιαλιστές. Για τις άδειες θα πρέπει να μπουν άμεσα στο αποθεματικό. Εάν επανεισέλθουν στην αγορά θα αποσταθεροποιηθεί ακόμη παραπάνω και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα το σύστημα εμπορία εκπομπών. Για το σύστημα ακύρωση θα ήθελα να προτείνω μία τροποποίηση στο κείμενο. Εάν έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια στο απόθυμα για διάστημα πάνω από δύο χρόνια, τότε το 20% θα πρέπει να διαγράφεται, να καταργείται μόνιμα. Ε, θα επανέλθω όμως στις τροπολογίες μου ε, σε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το σύστημα, για τα ανώτερα και κατώτερα όρια. Δεν βλέπω να συντρέχει λόγος να υπάρξουν σοβαρές τροποποίησεις. Ε, ίσως το κατώτερο όριο και ίσως η ετήσια προσαρμογή να ανέλθει στο 15%. Στις συζητήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Θεωρώ ότι είναι κατάλληλα τα όρια πάνω και κάτω από τα οποία αφαιρούμε ή ε, ξαμάζουμε στην αγορά ε, δικαιώματα εκπομπών. Η περίοδος των δύο ετών ε, θα ήθελα να είναι κατά τι μικρότερη. Η βιομηχανία ισχυρίζεται ότι δεν, μπορεί να, δεν έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή της ε, για το σχεδιασμό. Εγώ θα έλεγα ένα-ενάμιση χρόνο να ορίσουμε ως ανώτερη περίοδο, ούτως ώστε ε, να μπορούμε να παρακολουθούμε και τους κύκλους ε, της ύφεσης οικονομικής ανάπτυξης. Α, ναι, θέλω να κάνω και δύο ερωτήσεις στον κύριο Ταγιάννη. Στην τροπολογία 7 μιλάει για καθαρές ε, άδειες, ε, καθαρά δικαιώματα εκπομπών. Τι εννοεί ακριβώς, γιατί τα συζητούσε και με τους συναδέλφου από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και δεν καταλάβαμε. Για να τοποθετηθούμε υπέρ ή κατά, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει. Ε, και είναι και η άλλη. Η τροπολογία για την αεροπορία. 7. Τι εννοεί, ότι θα μπουν περισσότερα δικαιώματα στο αποθεματικό αν αποκλειστεί η αεροπορία από το σύστημα. Ευχαριστώ κύριο Σέριξον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα ότι το σύστημα ETS δεν λειτουργήσε ποτέ ε, όπως είχαμε προβλέψει. Το ξέρουν όλοι αυτό. Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί τώρα να το μεταρρυθμίσει το σύστημα, ώστε μακροπρόθεσμα να λειτουργήσει καλύτερα. Ε, είμαι υπέρ ε, του αποθεματικού ε, σταθεροποίησης αγοράς. Ο απότερος στόχος πρέπει να είναι να έχουμε εξελίξει προς μια σταθερότερη τιμή για τις εκπομπές διοξιδίου. Η βιομηχανία δεν κρίνει επίσης σημαντικό να μπορεί να υπολογίζει σε μια σταθερή τιμή για να κάνει και τις επενδύσεις της ε, προβλέποντας το μέλλον. Αν ακολουθήσουμε αυτό θα έχουμε εξάλλου και περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ενέργεια στην αγορά και άρα ε, αυτόματα χαμηλότερες τιμές ε, ενέργειας. Έτσι η βιομηχανία μπορεί να είναι όχι μόνο αποτελεσματικότερη αλλά και ανταγωνιστικότερη. θα έχουμε λιγότερες εισαγωγές επίσης και αυξημένη ενεργειακή ανεξαρτησία ε, που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό στόχος είναι σήμερα ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που θα έχουμε και λιγότερες εκπομπές διοξιδίου. Η τιμή των εκπομπών είναι προς συμφέρον της Ένωσης και της βιομηχανίας να παραμένει σε σταθερά επίπεδα και γι' αυτό Θεωρώ ότι είναι πλημελή η κατεύθυνση που ακολουθεί η πρόταση Ταγιάννη. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να τιμολογείται η, η εκπομπή. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τη μείωση των εκπομπών ούτε για την ε, αγορά και τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Νομίζω πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακολουθήσουμε αυτή τη σύσταση για άμεση ε, θέση σε ισχύ. Το νωρίτερο θα πρέπει να ήταν το 2019 19 μας λέει και το αργότερο 2021. Όχι, να σταματήσει το backloading τώρα και όλες οι άδειες αυτές να μπουν στο αποθεματικό σταθεροποίηση αγοράς. έτσι, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς μεγάλη διακύμανση των τιμών θα μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί ε, ομαλά το σύστημα. Και πολλά άλλα μπορούμε να κάνουμε για να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία, αλλά το σημαντικότερο ξαναλέω είναι άμεσα να αρχίσουμε να πάψει η λειτουργία του backloading και να αρχίσει να λειτουργεί το νέο αποθυματικό. Νομίζω στην Επιτροπή μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτή την συμβαστική λύση γιατί είναι ο σημαντικότερος στόχος από όλους. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ε, κύριε Έριξον, μιλήσατε ως, ε, με την ιδιότητα του σκιώδου εισηγητή από πλευρά ε, των Πρασίνων. Ο κύριος Λάμστορφ, αν κατάλαβα, θα μας μιλήσει από πλευρά της Γκουέ, τον κύριο Ένστ. Μάλιστα. Εμείς Πάντως έχουμε διαφορές ακόμη και στην ομάδα μας. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη και θα την επαναλάβω. Και μάλιστα ο Γέζι ε, διάσημος Πολωνός ε, συγγραφέας, το εξήγησε. Και ότι συμμετέχει κανείς σε ένα λαϊκό προσκύνημα με τεράστια προσέλευση δεν σημαίνει ότι δεν θα μυρίζει και τα πόδια των προσκυνητών. Οπότε το ίδιο ισχύει και για το σύστημα το εμπορίας εκπομπών που είναι το γενικό προσκύνημα. Ναι, μεν γενικό προσκύνημα, αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Υπήρχε η δυσοδεία των ποδιών. Και αυτό γιατί εισήχθη αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών και προσέθεσε στην ευρωπαϊκή αγορά ένα ακόμη στοιχείο κερδοσκοπίας και αβεβαιότητας. Το backloading, η αναβολή των δημοπρατήσεων των αδειών, έδωσε κάποια προσωρινή λύση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, γιατί αρχικά ο τόνος στοιχίζει 31 ευρώ και μετά την πτώση των τιμών ο τόνος στοιχίζει 6 με 7 ευρώ. Καταποντίστηκε η τιμή του άνθρακα το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι οι, κυρίως οι τραπεζικοί ε, ωφελήθηκαν και ενδιαφέρθηκαν για το backloading. Μερικοί τραπεζίτες ε, μου, έδωσαν, μου έθεσαν επιχειρήματα υπέρ του backloading, αυτής της αναβολής δημοκρατήσεων αδειών και είπαν ότι είναι υπέρ της ε, σταθερότητας του το κλίματος, αλλά άλλο έχω στο μυαλό τους. Ήθελαν ένα υποκατάστατο των παραγόγων. Γιατί κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, καταργήθηκαν ή περιορίστηκε η δυνατότητα επένδυσης ή ε, έκδοσης παραγόγων. Η δυνατοτητα επενδυσης σε εκδοσης παραγογων η προταση του κ. Ταγιάννη σίγουρα είναι καλύτερη από το προηγούμενο σύστημα του backloading, οπότε αυτός ο συμβασμός, αυτή η συμβαστική πρόταση είναι καλύτερη για την σύσταση αποθεματικού δηλαδή σταθερότητας αγοράς και θα πρέπει να την ε, εξετάσουμε διεξοδικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριο Σταμπουράνο από την EFDD. Συνάδελφος ε, Παξ ε, δεν θα παραμβεί και γι' αυτό το λόγο εγώ ομιλώ εξ ονοματός μου μόνο. Το θέμα είναι το εξής. Στην Ιταλία ακριβώς αυτή την εποχή υπάρχουν πολλές καταστροφές ας πούμε στην Τζένοβα, εκεί μιλάμε για τεράστιες υλικέ ζημιές και αυτό κάθε εβδομάδα. Σήμερα θα πλήξει πλημμύρα και τη Ρώμη. Ας μην ξεχνάμε και ότι κλείνουν μονάδες χάλιβα λόγω του ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός ακριβώς λόγω του συστήματος ETS. Γιατί παρεμβαίνω για τον εξής λόγο. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί. Όπως δεν λειτουργεί πια η παγκοσμιοποιημένη αγορά. Όσο πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το ελεύθερο παγκοσμιοποιημένο σύστημα, κανείς δεν μπορεί να μας σώσει και από το κλίμα και από ε, την απώλεια θέσεων απασχόλησης. Βεβαίως ε, η έλλειψη σταθερότητας είναι τραγική, είναι απογοητευτική. Εδώ έχουμε μια πρόταση, κάτι είναι και αυτό. Πρέπει όμως να επιτύχουμε πολλά περισσότερα και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτά που είπε ο κύριος Σταγιάννη εγώ τα στηρίζω ανυπερθέτως το σύστημα ETS και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δεσμευτούν να επενδύουν σε αυτό το σύστημα έτσι ώστε το, η παραγωγή να φτάσει σχεδόν στις μηδενικές εκπομπές. Νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστική σημασία. Όχι μόνο του 50%, εγώ θέλω και το 100% στο σύστημα ETS για να υπάρξει πραγματική αναδιάρθρωση και να μπορέσει να αποδώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. So we have finished... Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Λυπεί ο Για δύο λεπτά. Ο κύριος Γκερμπράντι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την διαρροή ε, άνθρακα, δηλαδή την κατάσταση των επιχειρήσεων. Με εντυπωσιάζει που το έθεσε ο κύριος Σταγιάννη, γιατί το γνωρίζει το θέμα καλύτερα από όλους μας. Ήταν μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ήδη ε, στην πρόταση για τη διαφυγή του άνθρακα μετά το 2020 φαίνεται ότι είχε λάβει υπόψη το, το αποθεματικό σταθερότητα αγορά. Και μάλιστα φαίνεται ότι υπήρχε πολιτική συμφωνία για 30 ευρώ τον τόνο για τον κατάλογο της διαφυγή του άνθρακα. Φαίνεται ότι δύο φορέ ε, έλαβε υπόψη τον υπολογισμό τη διαφύγη του άνθρακα ο κ. Σταγιάννη. Και αυτό είναι σαν να υπερβάλλουμε τη σημασία τη διαφύγη του άνθρακα. Παρόλο που εστερνίζομαι τι ανησυχίε ε, για το θέμα αυτό, θεωρώ ότι ήδη καλύφθηκε την πρώτη φορά. Ο βασικός σκοπός της σύσταση αποθεματικού σταθερότητα αγορά είναι να διορθωθούν οι αδυναμίε ε, του συστήματο εμπορία εκπομπών. Και γιατί θέλουμε να διορθώσουμε το σύστημα εμπορία εκπομπών. Καταρχήν δεν προσελκύσαμε τι επιχει... που επιθυμούσαμε για τι ε, καθαρέ τεχνολογίε. Και επίση ε, δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε του στόχου μα για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και και το θέμα του γενικού μα Οράματο για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Φυσικά θέλουμε να κρατήσουμε τι βιομηχανίε εντό της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Τι είδου όμω βιομηχανίε, τι βιομηχανίε του παρελθόντος ή νέε καινοτόμε βιομηχανίε του μέλλοντο. Ελπίζω το δεύτερο. Και μάλιστα σήμερα είχαμε στον Ολλανδικό τύπο το χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός Ολλανδού επιχειρηματία που ανέπτυξε δύο πρόσθετα για το τσιμέντο, γιατί η τσιμεντοβιομηχανία παράγει πολλά καυσαέρια. Χάρη στα δύο, αυτά συστατικά μειώνεται κατά 30% τα καυσαέρια λόγω του τσιμέντου. Και μάλιστα επιπλέον το τσιμέντο με τα δύο αυτά νέα συστατικά ήταν πολύ καλύτερη ποιότητα από το προηγούμενο σκυρόδεμα που χρησιμοποιούσαμε. Οπότε έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν ανώτερο που εκπέμπει πολύ λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Κάτι τέτοιο θέλουμε στην Ευρώπη και αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο εφόσον καταφέρουμε και ε, προσελκύσουμε αρκετές επενδύσεις στην καινοτομία. Και θα το, θα το επιτύχουμε μόνο με ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών που λειτουργεί εύρυθμα. Και όπως είπε ο κύριος Μίτς ε, στην προηγούμενη συζήτηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάθε χρόνο η Κίνα ε, επενδύει επιπλέον 22,5% στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και η Κορέα 5% ε, του ΑΕΠ της το επενδύει στην έρευνα και καινοτομία, ενώ η Ευρώπη μόνο το 2%. Συνεχίζουμε συνεχίσουμε τους ρυθμούς αυτούς θα μείνουμε σε χαμηλό επίπεδο. Ο κύριος Μαρτέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και κύριε Ταγιάννη που θέσατε επιτάπητο στο ζήτημα και ε, θέλουμε να μεριμνήσουμε για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Φυσικά με ενδιαφέρουν και εμένα τα θέματα των κλιματικών αλλαγών και της επανεκβιομηχανοποίησης, αλλά θα πρέπει να εντάξουμε τις βιομηχανίες σε ένα νέο κύκλο που θα είναι ένα άρετος κύκλος. Ας μην ξεχνούμε τους προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο του Κιώτο, καθώς και την περιβαλλοντική μας πολιτική. Θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας. Α μην ξεχνούμε αυτή τη σημαντική προτεραιότητα. Θα πρέπει όμω να διαφυλάξουμε και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μα. Να σταματήσουμε να είμαστε οι μεγάλοι αφελεί του πλανήτη, να επιβάλλουμε δρακόντια μέτρα στι δικέ μα επιχειρήσει και να, κλείνουμε, να κάνουμε τα στραβά μάτια για ό,τι συμβαίνει εκτό Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Φυσικά και οι επιχειρήσει θα μετεγκατασταθούν και θα παράγουν αλλού αυτά που θα πουλάνε στην Ευρώπη για να επανεντάξουμε τις επιχειρήσεις μας σε ένα νέο ενάρετο κύκλο θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε να επενδύσουν στις καθαρές τεχνολογίες. Και αυτό το απαγορεύουν οι κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε και ένα είδος διόρθωση στα σύνορα. Δηλαδή τα προϊόντα που προέρχονται έξωθεν και δεν σέβονται τις δικές μας προδιαγραφές και κανόνες θα πρέπει να αγοράζουν ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα από τις ενάρετε επιχειρήσει που θα επενδύουν σε φιλοπεριβαλλοντικές και καθαρέ τεχνολογίε. Μόνο έτσι με αυτού του είδου τα διορθωτικά μέτρα θα αποκαταστήσουμε έναν άρετο κύκλο. Γιατί ποιο είναι ο στόχο μα να διαφυλάξουμε τον πλανήτη. Αλλιώ, αν δεν το καταφέρουμε, πάντα θα υπάρχει ε, ένα μέρο όπου η ενέργεια θα είναι φθηνότερη και οι κανόνες για τη ρήπανση πιο ελαστικοί. Το θέμα είναι να ενθαρρύνουμε και τους υπόλοιπους αυτή τη υπόλοιπη υπήρου να μπουν σε έναν ενάρετο κύκλο όπω εμεί. Ο κ. Λεβαντόφσκι. Αυτό που θέλω να αναφέρω και να τονίσω είναι η δυσαναλογία, το δεν υπάρχει αντιστοιχεία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Κατά κανόνα λοιπόν στη λογική της αγοράς ε, ε, η τιμή είναι εκείνη που επαναφέρει την ισορροπία στην αγορά, αλλά σε αυτή την πρόταση όμως ε, δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία και γι' αυτό παρεμβαίνουμε. Υπάρχει και ένα δεύτερο μέτρο που προτείνεται, είναι το απόθεμα σταθερότητας και ο μηχανισμός αυτός. Ε, καταρχήν ε, έγινε λόγος για το backloading, 900 εκατομμύρια άδειες ε, και ποσοστώσεις. Μετά έγινε λόγος για τη σταθερότητα της αγοράς. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος έχει σχεδιαστεί. Εγώ προσωπικά θεωρώ τις ε, προτάσεις του κυρίου Ταγιάννη λογικές. Διότι ο κύριος Ταγιάννη τεχνητή καταδεικνύει ότι υπάρχει μια τεχνητή ισορροπία στο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών και αυτό δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός ούτε και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πώς θα ε, ισορροπήσουμε τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο εγώ στηρίζω τη σχετική τροπολογία που θίγει το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μας επανειλημμένως ταχθήκαμε υπέρ της επίγουσας εφαρμογής του θεματολογίου για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Γιατί η βιομηχανία θα γίνει ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας και θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, ποιοτικέ, ε, θα ενισχύσει τις, τις εξαγωγές και θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε καταπηγόντως όθηση στην απενεκβιομηχάνηση. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε φρέσκο χρήμα για τις επενδύσεις, για το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να γίνουν προσπάθειες επανεκβιομηχάνησης και να χρηματοδοτηθούν οι ενεργειακέ υποδομέ που είναι σημαντικό πυλώνας τη οικονομία. Όταν μιλούμε όμω για την βιομηχανία και το περιβάλλον φαίνεται να μιλούμε τελείω διαφορετικέ γλώσσε. Σημερίζομαι τις ανησυχίες του εισηγητή μα του κυρίου Ταγιάννη που λέει στο σχέδιο γνωμοδότηση ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε το στόχο μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με την ανάγκη προώθησης της βιομηχανίας μας. Οπότε η θέσπιση του αποθεματικού σταθερότητας αγοράς που με βρίσκει σύμφωνο θα πρέπει ε, αυτή η θέσπιση να γίνει υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ε, και τη θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη συγκυρία της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργοβόρου βιομηχανίας κυρίως. Προέρχομαι από το Ούλουγο που η βιομηχανία του αλουμινίου αντιπροσωπεύει το 30% του ΑΕΠ. Οπότε χαίρομαι που ο εισηγητής μας έχει επίγνωση της παρακμής της βιομηχανίας αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία των συνεπειών των ενεργειακών τιμών. Είναι θετικέ οι προτάσει του, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει ακόμη πιο φιλόδοξη. Και όχι μόνο να προτείνει το αποθεματικό σταθερότητα αγορά, αλλά και ένα φιλόδοξο και μεγαλόπνο σχέδιο για το ενεργειακό μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, γιατί αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μια και κάνουμε βήματα προς την φορολογική ένωση. Επιτρέψτε μια ακόμη φράση. Θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε στις ενεργειακές αλλαγές στην Ιφίλιο και να καταπολεμήσουμε ε, τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και για να γίνουμε πόλος καινοτομίας και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Έχουμε τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σταγιάννη επισημαίνεται πόσο σημαντικό είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και το να υπάρχει και ανάκαμψη της βιομηχανίας. Και λέει ότι μπορούμε να τα επιτύχουμε και τα δύο. Όμως ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτά είναι μια σαφής αντίφαση. Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής είναι εκείνο που αυξάνει το ενεργειακό κόστος και το ενεργειακό κόστος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, αποβιομηχάνηση στην Ευρώπη. Ο κύριος Σταγιάννη είπε ότι πρέπει να μειωθούν οι Εκπομπέ κατά 20%. Εκείνο που κάναμε όμω είναι δεν μειώσαμε τι εκπομπέ, αλλά τις πήγαμε αλλού, α πούμε στην Κίνα. Και με κάθε σεβασμό προ τον κύριο Γκεμπράντη, με την κατάσταση των εργοστασίων, ήδη λαμβάνει χώρα. Δεν είναι αν προβλέπουμε ή όχι, γίνεται. Και μεγάλε εταιρείε, όπω η Siemens, η BSF και άλλε κλείνουν τι μονάδε του και μετακινούνται ε, σε άλλα μέρη. Αυτό ήδη λαμβάνει χώρα και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίζεται. Εμεί ε, αντιμετωπίσαμε το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών σαν να ήταν μηχανισμός της αγοράς. Όμως, συνάδελφοι, αν χρειάζονται συνεχείς ρυθμιστικές παρεμβάσεις για να προσαρμόζεται η τιμή στην αγορά, αυτό δεν είναι μηχανισμός αγοράς, είναι αστείο. Ε, υπάρχει λοιπόν τώρα ε, μια ε, υστέρηση, έχουμε επίσης τις άδειε που συνδέονται με τη μετακατάσταση των επιχειρήσεων. Αυτά είναι παρανοϊκά κατά την άποψή μου. Στο δικό μας το κόμμα δεν μας αρέσει καθόλου η ιδέα της ε, νέας φορολόγησης. Όπως είπα όμως και κάποιοι σοβαροί οικονομολόγοι, αν θέλει κανείς να μειώσει τις εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, τότε ένας άμεσος φόρος θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός, πολύ πιο διαφανής και πιο καλός και για τη βιομηχανία. Γιατί λοιπόν στους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποτέ ότι απέτυχε ένα πρόγραμμα. Γιατί δεν κοιτάμε την αποτυχία κατάματα. Έχουμε το e system ETS, το ευρώ, μεγάλη αποτυχία και αυτό. Γιατί επιμένουμε να τα ε, στηρίζουμε αυτά τα προγράμματα και αυτούς τους μηχανισμούς όταν δεν αποδίδουν τίποτα. Ο κύριος Ρόιλ, επόμενος ομιλητής. Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να τσακώνεται, να διαφωνεί το τι είναι το σωστό και το τι όχι. Όμως αυτό που ισχύει είναι το εξής, ότι με, το, με την ε, εμπορία εκπομπών προσπαθούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και νομίζω ότι μέχρι τώρα λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Μειώθηκαν οι εκπομπές. Η Ευρώπη δεν τα πάει και τόσο άσχημα, παρότι, παρόλα αυτά όμως θέλουμε να παρέμβουμε το backloading και τώρα ε, να παρέμβουμε και πάλι με ένα ε, μηχανισμό ένα αποθεματικό. Ε, λέω λοιπόν στον κύριο Τεγιάννη το Προσέξτε, πόσο θα προχωρήσετε, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί κανεί ε, ένα στόχο με μεγάλο ενθουσιασμό, να θέλει δηλαδή να βελτιώνει την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Από την άλλη όμω να δυσκολεύει την κατάσταση βιομηχανία που είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Ήρθε λοιπόν η στιγμή εδώ στην Επιτροπή μα να αποφασίσουμε είμαστε υπέρ τη βιομηχανία ή όχι. Ε, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσει που θα κάνουν δύσκολο απασχολεί τη ζωή τη βιομηχανία, ή όχι συχνά το έχουμε συζητήσει, αλλά τώρα θα φανεί με την απόφασή μας το τι θέλουμε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πολλοί επιθυμούν προφανώς εξυγχρονισμό αυτού του συστήματος των εκπομπών, αλλά κύριε Ταγιάννη να έχουμε πάντα κατά νου τις επιπτώσεις, γιατί τελειώς είμαστε ανεύθυνοι. Και τέλος, κάποιος συνάδελφος είπε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε εκείνες βιομηχανίες που είναι καινοτόμες και όχι τις άλλες τις παλιές. Μάλλον δεν έχει καταλάβει. Η παλιά βιομηχανία που την ξέρω εγώ είναι πολύ εξ εξυγχρονισμένη, πολύ καινοτόμα, ε, συνεχίζει να εξυγχρονίζεται. Αυτό τώρα είναι ανοησία να λέει κανείς, η μένη είναι καινοτόμη και άλλοι δεν είναι. Ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ πολύ σύντομα να προσθέσω ότι εντάξει, πρώτα πρόταση του κύριου Ταγιάννη καλή είναι να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα επίσης με δεσμευτικές ρυθμίσεις, καλός και αυτός ε, και να μην υπάρχει προσμέτρηση κόστους ε, σε βιομηχανίες που κινδυνεύουν. Όμως, να πούμε το εξής, αυτό είναι συμβασμός και όλα τα άλλα που προτείνει ο κύριος Ταγιάννη, ας πούμε με το αποθεματικό που θα μειούται, αυτά είναι υπερβολικά για μένα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα της αγοράς που το έχουμε ήδη υπονομεύσει δύο φορές. Μία με το σύστημα και τώρα με το αποθεματικό. Κάθε μήνα κάνουμε και κάτι άλλο. Και απ' την άλλη μας ξεχνάμε ότι η βιομηχανία επενδύει με ορίζοντα 30 ετών. Ε, δεν γίνεται αυτό. Άρα δηλαδή πρέπει κάτι να κάνουμε και εδώ με αυτό το σύστημα που υπονομεύουμε την αγορά έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ρήγμα εμπιστοσύνη. Και αυτό που προτείνει τώρα ο κ. Σταγιάννη είναι ένα μπάλωμα θα το χαρακτήριζα. Είναι συμβιβασμό, δεν είναι εκείνο που εμείς ως ΕΛΚ είχαμε φανταστεί. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω το εξή στον εισηγητή μας. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εκφράζεται η άποψη ότι ε, θα μπορούσε κανείς να εγκρίνει τη δική του την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και με αυτή να πάνε ή να πάμε στις ε, διαπραγματεύσεις. Και εμείς ως Επιτροπή Βιομηχανίας θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να περάσει τουλάχιστον αυτός ο συμβασμός. Δηλαδή να μην εξαφανιστούμε εμείς τελείως ως Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ συνάδελφε πολύ σημαντικό και χρήσιμο να ακούμε τα προβλήματα από τη Σκοπιά και των δύο επιτροπών. Ο κύριο Γκέρεκ. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με το σύστημα εμπόριας εκπομπών και θεωρώ ότι από την αρχή ήταν αποτυχημένο το σύστημα. Και πραγματικά δεν έχει και μέλλον. Θα πρέπει να το βελτιώσουμε, αλλά ακόμη και να το βελτιώσουμε πάλι θα ανακύψουν προβλήματα αναποτελεσματικότητας. Τώρα, ποιο είναι το καθήκον μας. Εμείς θέλουμε να συνδέσουμε κάτι που παρουσιάζουμε πολύ θετικά, την ανταγωνιστικότητα με διασταλτική ερμηνεία και την εξαρτούμε την ανταγωνιστικότητα μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων με το θέμα της διαφυγής του άνθρακα. Μιλούμε ότι υπολογίζουμε σε 400 εκατομμύρια τόνους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το αποτυχημένο σύστημα που δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές του, των εκπομπών, για παράδειγμα των εκπομπών της δασοκομείας ή της γεωργίας, θα πρέπει το σύστημα αυτό λοιπόν να το καταργήσουμε όλος χερός και να στηριχθούμε σε ένα άλλο σύστημα. Για παράδειγμα, στο backloading, την αναβολή της δημοπράτησης των αδειών. Να συνδέσουμε το backloading με την αποτελεσματικότητα. Γιατί μόνο με την αποτελεσματικότητα θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και την καινοτομία και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ριζοσπαστικοί, να αν, αν κοπτόμαστε για τη σταθερότητα, νομίζω ότι θα την επιτύχουμε με την κατάργηση του συστήματο εμπορία εκπομπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να κάνω κάποιε παρατηρήσει συγκεκριμένα. Πρώτον, η Κομισιόν προτείνει την εισαγωγή αυτού του αποθέματος ε, για τη σταθερότητα τη αγορά μέχρι το 2020-2021. Εγώ προτείνω να γίνει πιο γρήγορα, το 2017. Και αυτό για ποιο λόγο. Για να δώσουμε ασφάλεια επενδύσεων στις επιχειρήσεις. Δεύτερον, όσον αφορά το backloading και τις άδειες που έχουν αποσυρθεί από την αγορά, αυτές να μην ξαναμπούν στην αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πλεόνασμα 2 δισεκατομμυρίων πιστοποιητικών αδειών. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταλήξει μια τιμή του 3,20. Αν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ουσιαστική ανταλλαγή εκπομπή, δεν θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα να πέφτει πιο κάτω η τιμή. Τρίτον, όσον αφορά ε, το χρόνο αντίδραση σε περίπτωση πλεονάσματος, να περιοριστεί. Τα δύο χρόνια είναι πάρα πολλά. Ε, και δεν φτάνει. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για να αντιδρούμε σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Τέταρτον, όσον αφορά την πρόταση Επιτροπής, εκεί πραγματικά πρόκειται απλά και μόνο για την εισαγωγή του αποθεματικού της εθερότητας της αγοράς και όχι για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Άλλο αυτό το δεύτερο. Και η Κομισιόν δεν αναφέρεται πουθενά στο εγγραφό της. Όσον αφορά την προστασία των ενεργοβόρων βιομηχανιών, πράγματι χρειαζόμαστε αποτελεσματικές ρυθμίσεις για μεταγκατάσταση επιχειρήσεων που θα πρέπει να λειτουργούν και μετά το 2020. Τώρα όμως το να γίνεται λόγος για την εισαγωγή αυτού του αποθεματικού, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλα τα άλλα. Πρέπει επίσης να λάβουμε μέτρα μετά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, γιατί και εκεί αναφέρεται ότι όσον αφορά το κλίμα και το ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να εγγυόμαστε την ανταγωνιστικότητα. Γίνεται λόγος για εγγύηση της, και διασφάλιση αν θέλετε της ε, ανταγωνιστικότητας ε, και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέω ο Τσανονάτο. Κοιτάξτε, έχουμε την προάσπιση του κλίματος ε, και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά να τα συνδυάσουμε με την διάσωση και ανάκαμψη της βιομηχανίας μας, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το σκεφτόμαστε σαν να είναι κάτι το πολύ απλό. Ε, είναι απολύτως απαραίτητο ε, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ε, να μετακινηθούμε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη του προβλήματος. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις αν το κάναμε θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ολέτριες συνέπειες. Άρα δηλαδή είναι απαραίτητο αυτά τα δύο στοιχεία να παραμείνουν συνδεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας από κοινού με διάσωση των βιομηχανιών και αυτό με βάση συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο Κιώτο. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα στοιχεία ως αντίθετα, τότε συμφωνώ με τον κύριο Ταγιάννη, τότε στην περίπτωση αυτή διαπράττουμε λάθος. Γιατί η πρόκληση είναι να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα στοιχεία να τα ε, διασφαλίσουμε από κοινού. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εγκαταλείψουμε απλά την ποσοτική προσέγγιση στη στάση μας και να περάσουμε ε, σε μία, να εγκαταλείψουμε την ποιοτική και να περάσουμε στην ποσοτική προσέγγιση. Η ποσότητα των φερμένων αριθμών του είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε και να κατανοήσουμε και πώς είναι συνδεμένα μεταξύ τους. Άρα δηλαδή κάτω από αυτό το πρίσμα μπορούμε να φτάσουμε σε μία λογική λύση. Και επίσης να σας πω και το εξής, εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε σαφή εικόνα του τι συμβαίνει ε, σε σχέση με την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και με την κατάσταση ή μετατόπιση δραστηριοτήτων που ε, παράγουν υψηλά ποσοστά διοξιδία του άνθρακα. Εγώ πιστεύω ότι επ' αυτού θα πρέπει να εμπαθύνουμε περισσότερο. Και θέλω να σας πω απλώς τη γνώμη μου και μετά ε, αφού έχουμε εμπαθύνει. Εδώ το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να ε, ανακτήσουμε ε, τα χρήματα, μάλλον τα έσοδα από το σύστημα ETS να τα επενδύουμε στην τεχνολογική έρευνα. Η κυρία Πιλάρ Δελκαστίο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα καινούριο. Θα ήθελα απλώς να πω ότι κατά τη γνώμη μου η πρόταση του κυρίου Ταγιάννη ευθυγραμμίζεται με αυτά που λέμε στην, στην Επιτροπή μας ε, για την ανάγκη διαφύλαξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Βέβαια η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει μια πιο παραδοσιακή στάση, αλλά και διαφέρεται περισσότερο για τις περιβαλλοντικές πτυχές. Είναι λογικό. Όταν συζητήσαμε το backloading, θυμάστε τις φοδρές αντιπαραθέσεις είχαμε και στην Επιτροπή Βιομηχανία, στην Επιτροπή μας. Διαφορετικά βλέπουν τα πράγματα οι δύο επιτροπές, η και η ΕΜΒΗ. Εμάς μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα συμφέροντα της βιομηχανίας και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της. Και είναι λογικό από τη στιγμή που είμαστε Επιτροπή Βιομηχανίας. Θα δούμε τώρα με τις τροπολογίες πώς θα τροποποιήσουμε την νομοδότηση. Πάντως ε, η πρόταση του κυρίου Ταγιάννη ευθυγραμμίζεται με τη δεδηλωμένη θέση της Επιτροπής Βιομηχανίας και Έρευνας. Σας ευχαριστώ. Ναι, θεωρούμε πως αυτό που μας υπεύθυνο γι' αυτό. Θα ζητήσω τον κύριο Ταγιάννη να συνοψίσει τη συζήτηση εφόσον ο εισηγητής μας θέλετε να προσθέσετε κάποιες παρατηρήσεις. Για τούτη, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και όλους εκείνους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο για να υπογραμμίσουν είτε την σύμφωνη είτε την αντίθετη γνώμη τους. Πάντως συμμετείχαν πάρα πολύ στη συζήτηση και αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους. Εγώ υπογράμμισα το θέμα του χρόνου. Όπως είπε και ο κύριο Μπράνκο, κατά την παρέμβασή του, οφείλουμε νομοθετώντας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως έχει σήμερα. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο ιδεατό. Όχι. Ζούμε σε ένα κόσμο που μαστίζεται από την κρίση. Υπάρχει πρόβλημα εκβιομηχάνη στην Ευρώπη. Υπάρχει πρόβλημα με τις ε, θέσεις απασχόλησης. Σας είπα, αυστριακές επιχειρήσεις ε, έφυγαν από την Ευρώπη και επενδύουν σε άλλα μέρη του κόσμου και πολλές άλλες. Για να μην αναφέρω και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση χάλιβα, παραδείγματος χάρη. Άρα δηλαδή ε, προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Αυτά είναι τα προβλήματα. Στην τροπολογία 15 προτείνω τον Ιούνιο του 2025 να αναθεωρήσουμε την κατάσταση. Τότε θα μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτά που εντωμεταξύ θα έχουν διαρματιστεί όχι το 2026 όπως αναφερόταν αρχικά, να κερδίσουμε ένα μισή χρόνο. Πιστεύω λοιπόν ότι πολλοί έχουν κατανοήσει ποιο είναι το πνεύμα που χαρακτηρίζει την πρόταση μου. Να υπάρχει ισορροπία. Αγώνας αφενός κατά της κλιματικής αλλαγής, από την άλλη όμως ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Όχι δηλαδή να επιβαίνει το κόστος για τις βιομηχανίες και το κόστος της ενέργειας που σήμερα για τις επιχειρήσεις είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που προκαλούν σημαντικά προβλήματα. Όσον αφορά τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 7, θέλω να είμαι σαφής από αυτού. Το κείμενο της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφές και γι' αυτό έγιναν αυτές οι προσθήκες. Και όταν προτείνω να αποκλείσουμε την αεροπλοεία, αυτό το λέω διότι με βάση δική μου την εμπειρία, επειδή ήμουν όπως ξέρετε επίτροπος μεταφορών και αργότερα επίτροπος ε, βιομηχανίας, θέλω να σας πω το εξή. Στην αεροναυπηγική οι εκπομπές δημιουργούν σύγχυση και δεν αφορούν την ε, ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανική. Υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείε που δεν είναι ευρωπαϊκές, γι' αυτό λοιπόν ε, αν αλλάζαμε τις ρυθμίσεις αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί βουλευτές είπαν ότι συμφωνούν με την άποψή μου, δηλαδή όλα τα κονδύλια που προβλέπονται για την αγορά του ETS να διοχετεύονται αυτά στην βιομηχανική ανάκαμψη. Θα ήταν ας πούμε λάθος να δοθούν για να μειωθεί αν θέλετε το δημόσιο χρέος και όχι για να ε, βρούμε μια λύση σχετικά με τις ποσοστώσεις. Αυτά που τα πληρώνουν οι βιομηχανίες σε τελική ανάλυση για να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Εγώ όταν ήμουνα επίτροπος είχα οργανώσει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μιλάγαμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ε, η βιομηχανία από μόνη της δεν είναι καθαρή αλλά για να είναι πιο καθαρή πρέπει να επενδύσουμε. 150 δις ε, του κοινωνικού προπλογισμού έχει αποφασιστεί να επενδεθούν στη βιομηχανία και τα 40 ε, αφορούν τον ορίζοντα του 2020 την έρευνα και την τεχνολογία. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Εγώ αυτήν είχα όταν ήμουν επίτροπος και σήμερα που είμαι ευρωβουλευτής, ναι στη βιομηχανία, αλλά να είναι σύγχρονη, όχι με τις υψικαμίνους που βγάζουν καπνό. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι, να γίνουν όλα αυτά βέβαια σιγά σιγά, γιατί αν ζητήσουμε ε, αν δεν έχουμε εφικτούς στόχους θα καταστρέψουμε τη βιομηχανία και θα δημιουργήσουμε και μεγάλο πρόβλημα στην, στις, ε, στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, θα γίνει οι επιχειρήσεις θα πάνε στην Κίνα που ήδη υπάρχει πρόβλημα ρήπανσης και εκεί θα αυξηθεί περισσότερο το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίσατε το λόγο. Ήταν πολύ πλούσια η συζήτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα συμφωνήσω με αυτούς που είπαν ότι η δυναμική από πολιτική σκοπιά που έχει δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο με πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Πέραν αυτού είχαμε ε, σε σχέση με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ και της Κίνα για την ε, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και μπορούμε λοιπόν και εμείς να ε, προωθήσουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές διοξιδίου. Για την πρόταση αυτή θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αφιερώσουμε δύο λεπτά στο στόχο αυτή τη πρότασης. Ίσως βοηθήσει στη συζήτηση. Αυτό το επιθυματικό σταθερότητα τη αγορά θα ε, καλύψει την υπερβολική προσφορά και θα καταστήσει επίση πιο ανθεκτικό το σύστημα ε, σε σχέση με μελλοντικά προβλήματα. Είναι μελλοντοστραφές ε, το σύστημα που προτείνουμε. Θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και θα ε, επικρατήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά. Εάν εγκριθεί η πρόταση εγκαίρως, δεν θα χάσουμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες για μείωση και σταθεροποίηση του κόστους, αλλά και για περισσότερες επενδύσεις σε αποτελεσματικότερες τεχνολογίες που μειώνουν την ε, κατανάλωση ε, του άνθρακα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που ίσως για κάποιους είναι αυτονόητο, αλλά είναι σημαντικό για την Επιτροπή, θα είναι αυτός ο μηχανισμός ένα χρήσιμο εργαλείο, διότι προσωρινά μπορεί να αυξήσει και τη ζήτηση σε περίπτωση που κρίνουν ότι ε, ελοχεύει ένας κίνδυνος ε, από πλευράς της ε, βιομηχανίας. Δηλαδή είναι αμφίδρομο το σύστημα και καλύπτει και την υπερβολική προσφορά αλλά και την υπερβολική ζήτηση. Για τη βιομηχανία επίσης ε, αντιμετωπίζει το θέμα της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων και αυτό αναφέρθηκε πολλές φορές στη συζήτηση, το τονίζω και εγώ, ότι η τωρινή τρέχουσα προστασία παρατείνεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ε, και πιστεύω ότι με αυτή την προστασία κατά της διαρροής ε, άνθρακα και με την δωρεάν προσφορά δικαιωμάτων εκπομπών είναι δύο κινήσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που τις χρειαζόμαστε προς το παρόν και άρα υπερασπιζόμαστε αυτό το σύστημα που θα σταματήσει κάποια στιγμή να ισχύει. Για το θέμα της διαρροής του άνθρακα, όπως είπε ο Επίτροπός μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα προετοιμάσουμε μια πρόταση που εξυπακούνται θα λαμβάνει υπόψη τα απορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εξάλλου το είπε και ο εισηγητής στην αρχή της συζήτησης ότι δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση ήταν ε, ε, σημαντικό ζήτημα αυτό της διαρροής του άνθρακα και θα ληφθεί αυτό υπόψη όταν προετοιμάσει η Επιτροπή την πρότασή της. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που προέκυψαν από τη σημερινή συζήτηση. Η μεταφορά των ε, αδειών από το σύστημα backloading στο νέο αποθεματικό, όπως είπε ο κ. Καλνιέτε, Δεν πρόκειται εμεί να εμποδίσουμε τέτοιε αλλαγέ εάν ε, συμφωνήσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Τέταρτον, ο χρονισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ταχύτερο δυνατόν να εγκριθεί αυτή η πρόταση, Πρόεδρε. για να διευκολύνουμε την έγκριση σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και τέλος, Όπως είπε και ο κύριος Καλνιέτε, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, θα εκπονήσει την πρόταση μεταρρύθμισης του ETS η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την προβλεψιμότητα στον βιομηχανικό τομέα. διότι εκεί θα προτείνουμε συγκεκριμένε αλλαγές για το σύστημα ε, μέχρι το 2030. Σας ευχαριστούμε. Όπως ε, λέγαμε και νωρίτερα συνάδελφοι, μπορούμε να ε, προσδοκούμε ευρία υποστήριξη για την πρόταση του εισηγητή μας. Ήδη το ακούσαμε από πολλούς συναδέλφους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για τη συζήτηση των συναδέλφων που τυχώς θα διαφωνήσουν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, ως συνήθω δηλαδή. Χαίρομαι λοιπόν που Ιβο Μπελέτ που είναι ο συγητής από την Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Μπέλετ ακούσατε όλες τις παρατηρήσεις, όλες τις προσδοκίες που έχουμε Και φαντάζομαι ότι σε κάποιο ορισμένο βαθμό τα είναι διαφορετική η συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα βρούμε κάποια συμβαστική λύση, τουλάχιστον στη δική μας συζήτηση έτυχε ευρεία υποστήριξη η έκθεση του κυρίου Ταγιάννη. Ήβο, μήπως θα ήθελες να πεις και εσύ κάποια πράγματα, παρακαλώ. This is the committee of είναι η Επιτροπή <laughs> Βιομηχανίας και Καινοτομίας και δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ε, δέκα χρόνια ήμουν εδώ στην Επιτροπή και την ξέρω πολύ καλά την Επιτροπή. Βλέπω πολλά οικία πρόσωπα. Τώρα είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σύντομα θα παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσής μου. Αυτό που κατάλαβα τώρα τη βάση της έκθεσης του Αντώνιο είναι ότι το σύστημα όπως έχει τώρα πρέπει να διορθωθεί. Νομίζω υπάρχει συνένεση σε σχέση με αυτό. Δεν υπάρχει ακόμη, αν κατάλαβα καλά, συνένεση για την ημερομηνία ε, έναρξης ισχύω. Ε, ε, υπάρχει το θέμα των αδειών που έχουν αποσυρθεί προσωρινά, για τις οποίες έχει αναβληθεί η δημοκράτηση. Πρέπει να επιληφθούμε και αυτού του ζητήματος. Το αποθεματικό σταθερότητα αγορά, όπω είπε και η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, δεν είναι νέα μορφή τη αναβολή δημοπράτηση του backloading. Αυτό ήταν προσωρινή λύση για να καλυφθεί η υπερβολική προσφορά. Το Κοινοβούλιο, όταν υποστηρίξαμε το backloading, ξεκάθαρα Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ε, διαρθρωτικού ε, χαρακτήρα μεταρρυθμιστική πρόταση. Αυτό κάνουμε τώρα, δηλαδή μεταρρυθμίζουμε το σύστημα της αγοράς ώστε να μην χρειάζεται πλέον αυτή η έκτακτη παρέμβαση, να αυτορυθμίζεται η αγορά αν θέλετε. Άκουσα πάρα πολλές επικοδομητικές προτάσεις. Είμαστε πολύ ανοιχτοί για να βρεθεί συμβαστική λύση σε συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανία για την πρόταση μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως πρότεινε και ο Επίτροπος Καλνιέται την περασμένη εβδομάδα, ελπίζουμε το Φεβρουάριο ή το Μάρτι να έχει βρεθεί ε, συμβαστική λύση και το ταχύτερο δυνατόν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πρώτα σας ευχαριστούμε συνάδελφε για τις παρατηρήσεις. Η καταληκτική η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι 24 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, στις 12. 12. Το έχετε όλοι το χρονοδιάγραμμα. Σε, μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να έχουμε όλοι καταθέσει τις τροπολογίες μας. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον εισηγητή μα τον εισηγητή από την ΕΜΒΗ, του ε, τους Σκιώδη, όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. 7. Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μισών επιχειρήσεων κατάσταση προόδου όσον αφορά την υλοποίηση παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούλβια Ραφαέλη, αναπληρώτρια τμήματάρχης της μονάδας επιχειρηματικότητας. Αυτό το πρόγραμμα ε, υιοθετήθηκε στα τέλη του 2013. Ο στόχος είναι να περιοριστούν τα προβλήματα ε, χορήγησης πίστης, χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκατό χιλιάδες επιχειρήσεις μπορούσαν να πάρουν χαμηλό το καδάνι από ένα αντίστοιχο με το κόσμο πρόγραμμα την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα, ήταν για την έρευνα και την καινοτομία, τώρα έχουμε το κόσμο και αρχίζει η συζήτηση. Μία ώρα έχουμε προβλέψει για τη συζήτηση, έχουμε ψηλοαργήσει. Μπορείτε να μην υπερβείτε τα 10 λεπτά, αν, μπορείτε. So, thank Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τους στόχους του προγράμματος COSME. Όπως είπατε αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το πρώτο πρόγραμμα που αφιερώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θεωρούμε ότι είναι από τους βασικούς μηχανισμούς και τα εργαλεία που θα έχουμε για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία τα προβλήματα και το διακύβευμα του κόσμου. Καταρχήν, τι δυσκολίες καλείται να, να διορθώσει το κόσμο μεταξύ 70 και 88% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν διοικητικές δυσκολίες, ε, κάτι που τους προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί τους αποτρέπει πολλές φορές από την ενασχόληση με το διασυνοριακό εμπόριο. Υπάρχουν χάσματα, κατακαιρματισμό, αποσπασματοποίηση και υπερβολική γραφειοκρατία στην εσωτερική αγορά, κάτι που εμποδίζει του πολίτε, του καταναλωτέ και τι μικρομεσαίε κυρίω επιχειρήσει να απολαύσουν των πλεονεκτημάτων τη εσωτερική αγορά. Είναι σημαντικό λοιπόν να δράσουμε για να αποφύγουμε περιττή γραφειοκρατία και τέτοια γραφειοκρατικά εμπόδια, αφήνοντα πιο ελεύθερο το δρόμο προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ένα άλλο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το σχετικά χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη. Όπω φαίνεται και στο Ευρωβαρόμετρο του 2012, μόνο το 37% των Ευρωπαίων πολιτών ε, θα ήθελα να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ενώ 51% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στις Ηνωμένε Πολιτείε και 56% στην Κίνα. Των πολιτών δηλαδή που θα ενδιαφέρονταν για αυτοαπασχόληση. Ο νέος δανεισμός σε επιχειρήσεις για χαμηλά ποσά κάτω του 1 εκατομμυρίου έχει μειωθεί κατά 40% στην Ευρωζώνη μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007. Επίσης παρατηρήσαμε ευθύνουσες τάσεις στην Ευρωζώνη, γιατί οι τράπεζες έγιναν πιο αυστηρές στο δανεισμό. Η πρόσβαση όμως στη χρηματοδότηση και στο δανεισμό είναι το πιο σημαντικό μέλημα των περισσότερων επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στο δανεισμό είναι το πιο φλέγον ζήτημα για τις επιχειρήσεις της Σλοβενίας, Ελλάδας και Κύπρου κυρίως. Και οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι πιο καινοτόμε επιχειρήσεις είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα για να βρουν χρηματοδότηση. Είναι εξωσημείωτη ότι η περιορισμένη διεθνοποίηση, δηλαδή οι διασυνοριακές δραστηριότητες τους εντός και εκτός της Ευρώπης ε, επηρεάζει τις επιχειρήσεις αυτές. Με βάση κάποιες εκτιμήσεις επί του παρόντος μόνο 25% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξάγουν ή κάποια στιγμή στη δραστηριότητά τους στην τελευταία τριετία είχαν κάνει εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το 13% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν τακτικές εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο 2% εξαγωγές εκτός της, ε, της χώρας εγκατάστασής τους. Ποιοι είναι τώρα οι στόχοι του προγράμματος COSME και πώς θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς. Το COSME, όπως είπα, είναι το πρώτο πρόγραμμα που αφιερώνεται ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να προωθηθούν οι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του και να τονωθεί η ανάπτυξή του. Επίση, στηρίζεται σε τοπικού ε, μεσάζοντε ε, και ε, τράπεζες, εμπορικά επιμελητήρια και πολλού τοπικού και εθνικούς φορεί που δρούν ω πολλαπλασιαστές. Επίσης, ο προπολογισμό είναι 2,3 δισεκατομμύρια για τη συνολική περίοδο εφαρμογής 2014-2020 έχει ετήσια προγράμματα εργασίας στο κόσμο και για το 2014 το πρόγραμμα εργασιών έχει προϋπολογισμό 246 εκατομμύρια. 246 εκατομμύρια προϋπολογισμό για φέτος. 20% του συνολικού προϋπολογισμού που προβλέπει ο κανονισμός προορίζεται για τη, βελτίωση της πρόσβασης, για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά. Για το 2014 είναι γύρω στα 61 εκατομμύρια που αφιερώνονται στο σκοπό αυτό. Οι δύο γενικότεροι στόχοι είναι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές και τις α, κοινοτικές και τις εξοκοινοτικές και η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο βασικός άξονας που χρηματοδοτείται από τους στόχους αυτούς είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων το δίκτυο αυτό συνεχίζει τις δραστηριότητες του προηγουμένου προγράμματος EIP και πραγματικά δίνει προστιθέμενη αξία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί είναι πραγματικά one-stop shop, μόνο απευθυντική θηρίδα στην οποία μπορούν να αποταθούν οι επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και έχει περίπου 600 φορείς στήριξη επιχειρήσεων σε πολλές χώρες ε, και το Μαρόκο, Αίγυπτο, Ισραήλ, την Ισία. Και στο μέλλον το δίκτυο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ε, και για άλλα κοινοτικά προγράμματα όπως το Horizon 2020 και θα παρέχει συμβουλές εθαρρύνοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν μέρος και σε άλλα κοινοτικά προγράμματα προκειμένου να αξιοποιηθούν οι συνέργειες των διαφόρων προγραμμάτων. από τα οποία μπορούν να αποφεληθούν οι, Ευρωπα... οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα η σχετική πρόταση δημοσιεύθηκε το Φεβράριο του 2014 και θα ενισχύσει τη στρατηγική υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο μέλλον. Και μάλιστα είχαμε πολλές προτάσεις με πάνω από 600 ε, οργανώσεις Η τελική υπογραφή για την παροχή επιχορηγήσεων θα γίνει το Φεβρουάριο του 2015 και ο δεύτερος διαγωνισμός ε, ανά, ε, αφορά γεωγραφικές ε, ζώνες που δεν καλύπτονται από τον πρώτο γύρο. Άλλη σημαντική πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από τους στόχους του κόσμου είναι οι διαδικτυακές πύλες. Εδώ έχουμε γνωστές πρωτοβουλίες όπως το Your Europe Business Portal το, η δικτυακή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το help desk για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κίνα, η Λατινική Αμερική και η ε, Νότια Ασία επίσης έχουν αντίστοιχα help desk που δίνουν άμεσα συμβουλές στις επιχειρήσεις ε, χάρη σε εμπειρογνώμονες ε, που δίνουν online τις πληροφορίες τους. Επίσης καλύπτουμε χώρες και περιοχές και δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένες αγορές που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ως προς τα IPR. Μάλιστα παρέχουμε υπηρεσίε και επιτόπου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη χώρα και γενικώ στην Ευρώπη, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν πριν να ε, ε, ξεκινήσουν να δραστηριοποιηθούν σε άλλες χώρες. Οι διάφορες προτάσεις ε, για τις ε, πλέον διαδικτυακές πύλες εξετάζονται και θα γίνουν λειτουργικές από το πρώτο τρίμηνο του 2015. 11% του προγράμματος COSME αφιερώνεται στη βελτίωση των, ε, του πλαίσιου εργασιών, του πλαίσιου συνθηκών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Και εδώ έχουμε δύο είδων δράσεις. Αφενός έχουμε δράσεις επιτόπου για να στηρίξουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εσωτερικές συζητήσεις για τη βιομηχανική πολιτική και τη πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ για παράδειγμα έχουμε δράσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της ομάδας Stoiber όπως λέγεται ή έχουμε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των, των πολιτικών εθνών. Επίσης έχουμε μια δεύτερη ομάδα δράσεων που είναι δράσεις που βελτιώνουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων τομέων. Εδώ συναντούμε πολλές διαφορετικές δράσεις για να στηριχθούν τα clusters, κάποιοι θύλακες ή άλλοι τομείς. Το 2014 ξεκινήσει μια δράση για τα δύο δράσεις για τα clusters, το πρόγραμμα αριστείας για τα clusters και η διεθνοποίηση των clusters. Τώρα για το, τον τομέα τουρίμ για τον τουριστικό τομέα. Ήδη το 2014 προκηρύξαμε διαγωνισμό για δράσεις που θα βελτιώσουν τις ε, διεθνείς τουριστικές ροές και τις ευρωπαϊκές τουριστικές ροές ε, και την ε, εποχική απασχόληση νέων στον τουρισμό. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε τη διαφοροποίηση της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα του τουρισμού. Ο τρίτος τομέας του κόσμου, εκεί έχουμε το 2,5% του συνολικού προπλογισμού και έχει ως στόχο να προάγει την επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν τα πιο δημοφιλή προγράμματα που χρηματοδοτούμε είναι το πρόγραμμα Έρασμος για τους νέους. Το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για να διευκολύνει προγράμματα κινητικότητας ε, για νέους επιχειρηματίες για να έχουν περισσότερες δυνατότητες ε, ε, να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες και επίσης και για να βελτιωθούν τεχνολογικές τους ικανότητες. Το 2014 εισαγάγαμε έναν άλλο κύκλο για την κινητικότητα και θα ξεκινήσει αυτό στην 1η Φεβρουαρίου του 2015 για μια περίοδο 24 μηνών. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 να έχουμε επιτύχει 1.300 ανταλλαγές με πάνω από 200 καταχωρισμένους επιχειρηματίες και με πολλούς ε, διαμεσολαβητές. Τώρα, το υπόλοιπο 60% ε, του προπολογισμού ε, για αυτό το ποσοστό θα δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου για να σας ενημερώσει πώς ακριβώς λειτουργούμε. Όπως ακούσατε ήδη προηγουμένως υπάρχει σημαντική και ριζική μείωση λόγω του προπλογισμού, ε, λόγω της οικονομικής κρίσης. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε εκείνες τις μικρομεσαίες που αλλιώς δεν θα είχαν καμία χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει πρόβλημα με τη δανειοδότηση στις αγορές, ε, κυρίως για αυτές που δεν έχουν εγγυητικές επιστολές. Εμείς αυτές θέλουμε να στηρίξουμε. Και όσον αφορά το πρόγραμμα, προβλέπουμε να στηρίξουμε 330.000 επιχειρήσεις 25 δις θα δοθούν για τη χρηματοδότηση αυτών των μικρομεσαίων. Το πρόγραμμα COSME προβλέπει δύο διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, το ένα είναι το ε, μετοχικό κεφάλαιο, το ενυπόθηκο δάνειο μάλλον, το equity capital και το άλλο είναι η κανονική δανειοδότηση. Σήμερα ακούσαμε την εισήγηση για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το οποίο και αυτό συμβάλλει και προβλέπει αυτά τα δύο μεμονωμένα εργαλεία. Όσον αφορά τις εγγυήσεις δανείων, αυτή την δυνατότητα, οι επιχειρήσεις μπορούν με τον τρόπο αυτό ε, να έχουν και να δημιουργήσουν νέα χαρτοφυλάκια. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη δυνατότητα στο βαθμό που μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν καταφύγει στο παρελθόν σε παρόμοια χρηματοδότηση ακριβώς ε, λόγω του ότι όλη αυτή η διαδικασία συνδέεται με πάρα πολλούς κινδύνους. Όσον αφορά τώρα τα ενυπόθηκα δάνεια, πρόκειται για επενδύσεις ε, που γίνονται ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη φάση που επεκτείνονται και μπορούν να λάβουν και τη μορφή, αυτές οι επενδύσεις τη μορφή συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο. Η Επιτροπή λοιπόν έχει αναθέσει την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων ε, στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο στο Λουξεμβούργο που είναι τη θεατρική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ε, εξειδικεύεται στο να προσφέρει υποστήριξη στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Κομισιόν υπέγραψε μια σχετική συμφωνία τον Ιούλιο αυτού του έτους και στις αρχές Αυγούστου είχαμε και δύο ε, προσκλήσει ενδιαφέροντο. Ε, η μία εκδήλωση αφορούσε την πρώτη δυνατότητα χρηματοδότηση και η δεύτερη, όπω σας είπα, τη δυνατότητα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. 30 Σεπτεμβρίου του 2020 θα έκλεινε, έκλεισε η δυνατότητα συμμετοχής. Πάντως αυτά τα εργαλεία εξαρτώνται από τη ζήτηση, εξαρτώνται πάρα πολύ από την αρχή οποίο προλάβει, θα χρηματοδοτηθεί πρώτος. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε το πρόγραμμά μας να ε, εφαρμοστεί το συντομότερο το πρόγραμμα IIF. Μέσα από αυτό μπορεί κανείς να δει ε, κατά πόσον οι ενδιάμεσοι επιθυμούν να έχουν αυτό το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογραφεί ακόμα καμία συμφωνία. Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Έχουν ε, κατατεθεί μία σειρά αιτήσεων και επίσης ε, γνωρίζουμε από συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη ότι υπάρχουν ε, κάποιες αιτήσει που βρίσκονται στη φάση προετοιμασίας. Τώρα, από τη στιγμή που έχουν υπογραφεί αυτές οι συμφωνίες, ε, πώς μπορούν να ενημερωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν έχει ε, φτιάξει μία πύλη, ένα πόρταλ και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κανείς πληροφορίες ε, και μπορούν πάρα πολύ εύκολα και να ε, πλογηθούν εκεί οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι μεγάλες αλλά και οι μικρομεσαίες. Μπορεί κανείς να κλικάρει σε μία χώρα και μία εταιρεία βάζοντας διάφορα κριτήρια ανάλογα με το τι θέλει να χρηματοδοτήσει μπορεί να διαπιστώσει η εταιρεία μόνη της κατά πόσον υπάρχουν κοινωτικά κονδύλια για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, πέρα από τα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία. Οι υπόλοιπε ε, δραστηριότητες ε, ε, χρηματοδοτούνται από την Ιάσνα. Είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν και για φέτος και για την επόμενη χρονιά, το 2015, έχουν ήδη ληφθεί ε, κάποιες ε, αποφάσεις χρηματοδότησης, ε, λήφθησαν τον Οκτώβρη αυτού του έτους. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρουμε αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και για τις παρατηρήσεις σας που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για όλους μας για τις διαφάνειες που μας δείξατε, για τις ερμηνείες που δώσατε, για τις παρατηρήσεις σας. Λόπες Βερμέιο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ. Συμφωνούμε με την πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, όμως έχω εντοπίσει πολλές αντιφάσεις στην πρόταση. Για παράδειγμα, περιορισμός των κονδυλίων της πρωτοβουλίας. Όπως είπε το Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, το 2012 ε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα που δεν είχε διορθωθεί ακόμη. Δεύτερον, δεν ε, υπάρχει συντονισμός με τις άλλες προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωρίς πολιτικές για την τόνωση της ζήτησης ε, θα υποφέρουν από την αδυναμία διάθεση των προϊόντων τους. Χρειαζόμαστε μια πολιτική οικονομικής ανάπτυξης και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που θα καλύπτει τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχει ακριβώς ομοιομορφία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οπότε στρατηγικέ, όπως ο ορίζοντα 2020 δεν επαρκούν. Οι πολύ μικρε επιχειρήσει έχουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά και πολλά, πολλοί στόχοι όπω χρηματοδότηση, εξαγωγές κτλ. Φαίνεται ότι, να, φαίνεται ότι ε, σχεδιάστηκαν για τι μεγαλύτερε επιχειρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεκριμενοποιηθούν κάποιε προτάσει για να προσαρμοστούν στι ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Επίσης ε, και το πρόβλημα του δανεισμού που αφορά κυρίως την έλλειψη ζήτηση. Θα πρέπει τώρα ε, για το, τα κεφάλαια κινδύνου, αν έχουμε ποσοτικά στοιχεία, θα αποσταθεροποιήσουμε τις ε, παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ των τραπεζών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενώ η σχέση αυτή είναι σημαντική για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θέλουμε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, αλλά θέλουμε να προσαρμόσουμε τα υπάρχοντα εργαλεία στην ε, διαφορετικότητα και την πολυμορφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κρίμα που ε, δεν λαμβάνεται υπόψη στους στόχους συντόνωσης της αυτοαπασχόλησης, γιατί με το ε, μέτρο αυτό δυστυχώς ενισχύεται την ψεύδο απασχόληση και των ε, αυτοπασχολούμενων που εξαρτούνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις που καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα ή τα υπονομεύει ή τα υποβαθμίζει. Έτσι ενισχύεται η τα υπονομευει τα υποβαθμιζει ρητορική που φέρνει ανθρώπους ε, να αυτοπασχολούνται αλλά παρόλο αυτά να σχεδόν να μην έχουν μισθούς. Νομίζω ότι κάτι που λείπει από την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το να εστιαστεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κύριο Σκέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε ε, για την παρουσίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και είναι ζωτική σημασία να εστιαστούμε στους τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί πραγματική ανάπτυξη. Δηλαδή, ε, ανάπτυξη της μικρομεσαίας και όχι για τις πολυεθνικές. Συχνά ακούγεται η εξή ανησυχία ότι κάποιες μικρομεσαίες ε, διστάζουν και δεν θέλουν να έχουν συναλλαγές σε άλλες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός. Λόγω των διοικητικών δυσκολιών παραδείγματο χάρη ε, είναι ο βασικότερος φραγμός. Πώς θα υπερβούμε αυτό το εμπόδιο. Εάν ε, υπάρχουν κατά την αντίληψη των μικρομεσαίων διοικητική φραγμή στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούν λοιπόν να τις ξεφορτωθούν, πώς μπορούν να ε, επεκτείνουν τις δραστηριότητες Στη συνέχεια μιλήσατε για μείωση του διοικητικού άχθους πάλι για τις μικρομεσαίες. Έχει ποσοτικοποιηθεί, μπορείτε να μας πείτε τι εννοούν στην πράξη, ποιοι είναι αυτοί οι φραγμοί. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να το σάρουμε. Διότι όταν κανείς ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες δυσκολεύεται να βρει ικανοποιητικά στοιχεία. Στη συνέχεια πολύ χάρηκα που μιλήσατε για τα εμπορικά επιμελητήρια. Εάν θέλουμε να προβάλλουμε το κόσμο και να ξεκινήσει μια δυναμική για να δημιουργηθούν νέες μικρομεσές, τα εμπορικά επιμελητήρια που ε, δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς έχουν σημαντικότατο ρόλο να παίξουν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα σε επιχειρηματίες, ε, επιχειρήσεις που υπάρχουν, ή άλλες που ξεκινούν και εμάς. Τι έχετε προβλέψει για να εμπλακούν περισσότερο ε, τα βιομηχανικά επιμελητήρια σε αυτό που ουσιαστικά είναι η δουλειά τους. Σας ευχαριστούμε ε, για τις ερωτήσεις και για τις παρατηρήσεις σας. Κυρίες μου, θα μπορούσα να σας ζητήσω να δώσετε απαντήσεις. Good. Ευχαριστώ. Ε, για την προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις. Ναι, είναι πρόβλημα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ορισμένες φορές ε, δικαίως λέγεται ότι οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι αποφελείς για τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, γιατί οι μικρές δεν ξέρουν πού να βρουν αυτά που χρειάζονται. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του κόσμου είναι αποκλειστικά και μόνο για τις μικρομεσαίες. Μία επιχείρηση που δεν είναι μικρομεσαία δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τις χρηματοδοτήσει η τράπεζα, αλλά εάν είναι να δώσει ένα δάνειο και λέει ο ε, διαμεσολαβητής ότι θα φτιάξουμε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων για να υποστηρίξουμε μόνο τις μεταφορές, εάν υποστηρίξουμε μια τέτοια μεταφορά για μια όχι μικρομεσαία επιχείρηση, δεν μπορεί να έρθει αυτός ο διαμεσολαβητής και να βάλει το δάνειο αυτό στο δικό μας το χαρτοφυλάκιο του κόσμου θα έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια αντιεπιλεξιμότητας. Δηλαδή μόνο οι μικρομεσαίες θα υποστηρίζονται. Αυτό ισχύει και για το Equity Facility for Growth, το ειδικό εργαλείο του κόσμου που προωθεί τις επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης. Ε, όταν γίνεται η πρώτη επένδυση και είναι ε, κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, ή επειδή ένα ταμείο που ε, χρηματοδοτείται ε, από ένα τέτοιο management fund αλλά δεν είναι πλέον στην ε, εναρκτήρια φάση, στη φάση ανάπτυξη, συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη, αλλά αυτό δεν, το, το πρόβλημα είναι, το, μάλλον το κριτήριο είναι ότι πρέπει αρχικά να είναι μικρομεσαία και να προωθηθεί στην ανάπτυξή της. Για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε σχέση με την ε, παγκοσμιοποίηση, σας μίλησα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι τοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των εμπερικών επιμελητηρίων, ε, ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό απαντώ στο ερώτημά σας συμφωνώντας ουσιαστικά. Οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν την πραγματικότητα, ξέρουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μικρομεσαίων. Ε, το ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο κάνει σεμινάρια για τις επιχειρήσεις, αλλά όχι αυτό, δίνει πληροφορίες που ε, ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις για να προετοιμάσουν ε, τη χρηματοδότηση ή για να βγουν από τη χώρα. υπάρχει δικτυακή πύλη και IPR σελίδα ε, που δίνουν πληροφορίες σε επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν εκτός από τη χώρα τους. Επίσης, ε, για να βγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσουν συναλλαγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είναι πολύ καλά αυτά τα σημεία επαφής για ενημέρωση και θα λειτουργούν και ως σύνδεσμοι με τρίτες χώρες. Ο πρώτος προορισμός φυσικά για τις εξαγωγές είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το σημείο επαφής και να υπάρχει και ανταλλαγή έτσι, πληροφοριών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Θα θυμάστε επίσης πως ε, υπήρχαν διάφορες αποστολές αναπτυξιακές. Ο πρώην Αντιπρόεδρος Σταγιάννη ηγήθηκε πολλών τέτοιων δράσεων και πολλές τέτοιες δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα COSME. Για το άλλο ζήτημα, της μείωσης του διοικητικού άχθους, ε, το COSME είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε πληροφορίες ε, για την ε, αντιμετώπιση των ε, διοικητικών εμποδίων. Δηλαδή δεν είναι τα εντοπίζουμε μόνο τα εμπόδια, τα αντιμετωπίζουμε κιόλα. Προτείνουμε λύση. Ο κύριος Ζωρίνιο, πολύ ευχαριστώ πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό από οικονομικής πλευράς αλλά και από πλευράς ε, της εγκύτητας ε, ε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικότατους τομείς που αναφέρατε, η συνεργασία που είναι και ο σημαντικότερος, η ικανότητα ε, της δημιουργίας μιας κρίσιμης μάζας, ούτως ώστε αυτές οι μικρομεσαίες να μπορέσουν να εξάγουν είτε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά η χρηματοδότηση και τρίτον η διεθνοποίηση, η παγκοσμιοποίηση. Ε, ένα πρακτικό ερώτημα έχω που σχετίζεται με τον τρόπο που συνδυάζεται αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τα εθνικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε, στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πορτογαλία τουλάχιστον υπάρχουν παρεμφερεί προγράμματα σε ε, επίπεδο Πορτογαλίας, ε, πάνω κάτω ίδιες προϋποθέσεις, ίδιοι στόχοι. Αυτό το πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ε, υποστηρίζει επιχειρήσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν ομίλους. Αυτή είναι η διάσταση της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να συνεργαστούν επιχειρήσεις ιταλικές, πορτογαλικές, ισπανικές και να δημιουργήσουν έναν όμιλο. Μια κοινοπραξία. Τι γίνεται στην πράξη. Έχουμε ε, φάμιλα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Τι γίνεται λοιπόν Μπορεί να απορριφθεί μία επιχείρηση και μετά να πάει να καταθέσει την αίτηση στον κόσμο ε, ή αντίστροφα. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπληρωματικότητα με τα εθνικά προγράμματα και κατά πόσο αντίστοιχε πρωτοβουλίε έχουν αναλάβει και τα κράτη-μέλη. Το σημείο φετηρή είναι διαφορετικό. Υπάρχουν μεγάλε διαφορετικέ μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορέ στη χρηματοδότηση. Μερικέ χώρε χρησιμοποιούν εκτενώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε τοπικό και περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και άλλε ελάχιστα ή καθόλου. Ε, και ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει ότι τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να είναι συμπληρωματικά με τα εθνικά και τα τοπικά, όχι να τα υποκαθιστούν. Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Σε ό,τι αφορά το χρέος της εγγύησης και της αντιγγύησης όταν κάποιος υποβάλλει ένα αίτημα στο, στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και για νέε δραστηριότητε ή προϊόντα θα πρέπει καταρχήν να αποδείξει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το θέμα αυτό γιατί υπάρχει το στοιχείο του κινδύνου και επίσης ότι δεν μπορεί να ότι έχει ένα είδος κάλυψη από αλλού, ώστε εμείς να συμπληρώσουμε τη χρηματοδότηση. Αν μια χώρα είναι πολύ δραστήρια και έχει πολλά θέματα, ήδη πολλά, πολλές πρωτοβουλίες, τότε το top up, εκεί που συμπληρώνουμε εμείς, τσοντάρουμε στο, στα, στις κρατικές προσπάθειες, είναι ελάχιστα, γιατί θέλουμε το κόσμο να ενισχύσει κυρίως ε, πρωτοβουλίες ε, ε, σε τα θέματα αυτά. Αυτά για το χρέος. Σε ό,τι αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το equity, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για να στηρίξουμε κάποια κεφάλαια επενδυτικά, δίνουμε έμφαση στο διασυνοριακό χαρακτήρα. Γιατί μερικές φορές τα περιφερειακά προγράμματα ε, είναι τοπικώς ε, εστιασμένα σε συγκεκριμένη περιφέρεια. Δεν έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον διασυνοριακό χαρακτήρα, παρόλο που κάτι τέτοιο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο και γι' αυτό το αποφεύγουν κυρίως οι επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμε οι, οι παρατηρήσει συγγνώμη, και εξηγήσει που μας δώσατε. Γιατί γνωρίζουμε ότι το κόσμο είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Βρίσκεται στα σπάργανά του τώρα μόλις ξεκινά. Και περιμένουμε 340.000 δάνεια. Και αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία φάση είχαμε 100.000 μέσα σε μία πενταετία θα έχουμε τριπλάσιο αριθμό. Αν το συγκρίνετε με το προηγούμενο πρόγραμμα, είχαμε 340.000. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το αριθμό των δανείων, τις 340.000. Γιατί χάρη στην προσθετικότητα εμείς ε, δίνουμε χρηματοδοτική υποστήριξη για δάνεια που οι μεσάζοντες δεν θα είχαν από αλλού χρηματοδότηση. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε το ίδιο επίπεδο στήριξη με το προηγούμενο πρόγραμμα. Αν και αυτή τη φορά έχουμε περισσότερα κονδύλια. Αλλά ακριβώ οι συναλλαγές που καλύπτουμε έχουν μεγάλο παράγοντα κινδύνου. Σα ευχαριστώ λοιπόν και για τις παρατηρήσεις και για την παρουσίαση και τις εξηγήσει. Μας ενδιαφέρει πολύ στην Επιτροπή Ήτρε η πρόοδο του προγράμματο και η μεταξέλιξή του. Φτάνουμε τώρα αγαπητοί συνάδελφοι στο τελευταίο θέμα του προγράμματος ε, τη ημερήσια διάταξη, στο σημείο 8, την αποστολή αντιπροσωπή τη Επιτροπή ΣΥΤΡΕ στην ένατη συνεδρίαση του Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, 2 με 5 Σεπτεμβρίου 2014. Μετά αυτή παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας που έγινε στην Τινησία το 2005. Επικεφαλής της Αντιπροσωπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής για το πολύ αυτό σημαντικό θέμα, το ψηφιακό θεματολόγιο δηλαδή, την ενιαία αγορά και το καθεξής, είναι η κυρία Πιλάρ Δελκαστίγιο Βέρα. Στην εισηγητριά μας λοιπόν θα δώσω το λόγο για να μας κάνει την ενημέρωση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της διακυβέρνησης, του Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε όλοι κουρασμένοι, έχουμε περάσει ήδη αρκετές ώρες συνεδρίασης. Θα είμαι λοιπόν πολύ συνοπτική στην ενημέρωση και θα σας στείλω πιο διεξοδικές πληροφορίες ηλεκτρονικώς. Εδώ θα επικεντρωθώ στα ουσιώδη. τι διανύθη, ποια ήταν τα κύρια σημεία αυτού του Παγκόσμιου Φόρουμ για το διαδίκτυο που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Το Φόρουμ Διακυβέρνηση του Διαδικτύου είναι άμεση απόρρια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για το Διαδίκτυο που έγινε στην Τινησία το 2005. Βασικός ε, στόχος είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε ένα γενικό φόρουμ και να έχουν διάλογο για θέματα κρατικών πολιτικών με θέμα το διαδίκτυο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στο παρελθόν, θέλουμε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο φόρουμ αυτό. Εκπροσωπούμε την Επιτροπή Ήτρε, την Επιτροπή Πολιτισμού και τη ΣΤΟΑ. Δυστυχώς, ο συνήθως η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε μόνο λιγομελή αντιπροσωπεία για την συμμετοχή στο φόρουμ. Ήμασταν μόνο τέσσερις στην αντιπροσωπεία. Σε σχέση με το παρελθόν ήμασταν πολύ λιγότερο. Δύο εκπρόσωποι από την Ήτρε, η υποφαινομένη και ο Ρενάτο όρο από τους σοσιαλιστές. Η κυρία Βερχάιν ήταν από την Επιτροπή Πολιτισμών και ένα ευρωβουλευτή από την Επιτροπή στο Α. Σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις έχουμε ένα γενικό θέμα, ένα οριζόντιο θέμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και άλλα στην πορεία. Το γενικό θέμα της τελευταίας συνεδρίασης είναι, ήταν η σύνδεση των υπήρων για διευρυμένη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Οπότε, με βάση αυτό το γενικό πλαίσιο, είχαμε και επιμέρους θέματα που τα συζητήσαμε σε διάφορα, διάφορα εργαστήρια. Για παράδειγμα, η διακυβέρνηση του διαδικτύου μετά το 2014 και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στις αρχές του 2015 τα Ηνωμένα Έθνη θα τον να λάβουν μία απόφαση για το μέλλον των φόρα διακυβέρνησης του διαδικτύου, γιατί εδώ και 10 χρόνια είχαμε αυτό το θεσμό. Η γενική θέση και κρατούσα θέση στο φόρουμ ήταν υπέρ της συνέχισης τέτοιο, πρωτοβουλίας. Και μάλιστα πρότεινα και την αύξηση του προπολογισμού. γιατί είναι πενιχρά τα μέσα χρηματοδότηση του φόρουμ. Επίσης θέλουμε τη συμμετοχή όλο, όσο, όσο περισσότερο γίνεται ενδιαφερομένων στην διακυβέρνηση του διαδικτύου. Αυτό ήταν σημαντικό αίτημα της συζήτησης. Και εδώ και χρόνια γίνεται συζήτηση μεταξύ δύο θέσεων. Αφενός έχουμε την προσέγγιση την πολύπλευρη, της πολύπλευρης διακυβέρνησης του διαδικτύου. Έχουμε χώρες που είναι υπέρ μιας πιο διακυβερνητικής μεθόδου για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Αλλά στο ίδιο το φόρουμ διακυβέρνηση του διαδικτύου η κρατούσα άποψη είναι, ήταν της πολύπλευρης διακυβέρνησης του διαδικτύου. Multi-stakeholder. Επίσης και τα περιφερειακά και εθνικά φόρουμ διακυβέρνησης θα πρέπει να λάβουν μέρος με ανταλλαγή πρακτικών, το βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για θέματα όπως η ανάπτυξη πολύπλευρων μηχανισμών διακυβέρνησης, ρύθμιση και επίλυση του θέματος των ανεπιθυμήτων μηνυμάτων, των spam, ενίσχυση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και δημιουργία πρόσφορου κλίματος για την ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου και επίσης σημαντικά μέτρα προστασίας των παιδιών επιγραμμικά. Άλλα θέματα σημαντικά, η οδετερότητα του δικτύου, η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, βελτίωση πρόσβασης και ανάπτυξη του διαδικτύου, καθώς και ψηφιακή εμπιστοσύνη. Ή ένα μήνυμα προς τους νέους. Είχαμε επιμέρους εργαστήρια, όπως σας είπα. Η δική μας αντιπροσωπεία συμμετείχε επίσης σε μερικά από αυτά Ε, είχαμε ένα εργαστήριο με θέμα διαδίκτυο και θέσεις απασχόλησης. επικοδομητική ή αποκοδομητική δημιουργία. Ε, λογοδοσία στην πολύπλευρη διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση του ίντερνετ, προκλήσεις, θέματα, ρόλοι. Η περίπτωση μεταβλητής γεωμετρίας ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση ουδετερότητα, η εποχή του διαδικτύου, προσαρμογή στο, στην ατζέντα των νέων πνευματικών δικαιωμάτων, πολιτικές και πρακτικές ε, για να επιτρέψουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων, ανοιχτά δεδομένα και διακυβέρνηση έκδοση των δεδομένων ε, στην εποχή των μέγα δεδομένων η πρόθεση των δικαιωμάτων των νέων. Είχαμε συνεδριάσεις ε, και συναντήσεις με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών, ε, με εκπροσώπους δημοσίων αρχών και φυσικά πολλών χωρών. Είχαμε συνάντηση με την UNESCO με θέμα την ψηφιακή ασφάλεια των δημοσιογράφων. Είχαμε συναντήσεις με πολλούς οργανισμούς που ασχολούνται και οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Συναντηθήκαμε και με την αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα εκεί η Αμερικανική αντιπροσωπεία διατράνωσε την προτίμησή της για την πολύπλευρη μορφή διακυβέρνηση του διαδικτύου. Είναι αναφανδόν υπέρ της πολύπλευρης διακυβέρνησης του διαδικτύου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε εκπροσώπους από πάρα πολλές χώρες ε, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο. Και τέλος να σας αναφέρω κάμια δυο άλλες συναντήσεις που είχαμε, δεν θα τις αναφέρω εξαντλητικά, με την ICAN. Ήταν πολύ σημαντική η συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, η ICAN είναι ο συνεταιρισμός που αφορά την κατανομή των ε, ε, ονομάτων και ε, αριθμών. Και υπάρχει σύμβαση με τις ΗΠΑ για εξασφάλιση απόλυτης ανεξαρτησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα θέματα διακυβέρνησης του διαδικτύου. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση για την ICAN και την ΙΑΝΑ που επίσης εξαρτάται από την ICAN που όπως σας είπα είναι η αρμόδια αρχή το σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών. Τέλος, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ότι καταρτήσαμε και δημοσιεύσαμε κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας μας με τίτλο «Μάχη για ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο». Η κοινή δήλωση προσυπογράφηκε από την Έλλη Κρούς, την Αντιπρόεδρο και όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τονίζουμε στην κοινή αυτή δήλωση ότι η πρόσβαση στο ίντερνετ έχει κρίσιμη σημασία για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να έχουμε συνεχή πρόσβαση σε ανοιχτό και ελεύθερο ίντερνετ που είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Και φυσικά το θέμα της επιτήρησης ε, σε μεγάλο βαθμό μειώνει την εμπιστοσύνη στην διακυβέρνηση του διαδικτύου. Θα πρέπει η διακυβέρνηση να γίνει πιο διαφανή, διαφανής, ε, υπόλογη και να μην αποκλεί κανέναν. Στην Κωνσταντινούπολη έλαβε χώρα αυτό το φόρουμ και μετά τις ε, δράσεις της τουρκικής, ε, των τουρκικών αρχών να επιβάλλει λογοκρισία στα κοινωνικά μέντια, Είχαμε την περίπτωση φυλάκισης δημοσιογράφου και πολλές διαμαρτυρίες. Είπαμε ότι η περιορισμός των θεμελιωδών ελευθεριών, ε, όποια μορφή και αν έχει, είναι απαράδεκτος. Αυτά. Σας είπα, σύντομη θα είναι η ενημέρωση. Το είπα και το έκανα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, εκθεσή σας, για την παρουσίαση που κάνατε, για όλα αυτά τα σχόλια σχετικά με το μέλλον. Και θα ήθελα να την ε, παρακαθήμενή σας, αν θέλει και αυτή να προσθέσει κάτι. Νομίζω ότι η Πιλάρ Καστήλιο ανέφερε τα σημαντικότερα θέματα. Ε, αυτό που πραγματικά επικράτησε ήταν το θέμα του ε, IGF, ε, του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Ε, εδώ και αρκετά χρόνια πολλές χώρες αγωνίζονται να έχουν μια περισσότερο διακυβερνητική προσέγγιση. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε κατά το παρελθόν το θέμα του διαδικτύου είναι πολύ ικανοποιητικό, πολύ ισορροπημένη εκπροσώπηση του κλάδου της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών. Υπήρχε λοιπόν ε, πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εμείς ε, στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση πολλών και πολλαπλών ενδιαφερομένων. Είμαστε σαφείς επ' αυτού και επιθυμούμε να ανοίξει ο δρόμος για να ληφθεί μία απόφαση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να ε, δοθεί εντολή στο Φόρουμ Διακυβέρνησης Δικτύου για το μέλλον. Αυτό που έχει σημασία και θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας οποτεδήποτε ε, οργανώνουμε ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι το EuroDIC, είναι η ευρωπαϊκή εκδοχή του Φόρουμ Διακυβέρνηση Διαδικτύου. Υπάρχει μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα σε αυτά που συζητούνται στα εθνικά, στα ευρωπαϊκά, το EuroDIC και επίσης αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν και ε, χειροπιαστά συμπεράσματα για το μέλλον του IGF, του Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου. Όταν συνδυέται κανείς με ανθρώπους από άλλες υπήρες βλέπει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα επόμενα χρόνια για μένα που είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίες έκφρασης, ε, προστασίας παιδιών, δημοσιογραφία, αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ λοιπόν ε, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το Φόρουμ Διακυβέρνηση Δικτύου. Αλλά τα συζητήσαμε αυτά και συζητήσαμε γενικά στην Επιτροπή Πολιτισμού αν ε, στο μέλλον μπορούμε να στείλουμε δύο μέλη σε αυτό το Φόρουμ γιατί η Επιτροπή Πολιτισμού κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να στηρίξω την Πιλάρ. Ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ο ρόλος που μπορεί να ε, διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη μεταβατική φάση και στο μέλλον της ICAN. Νομίζω η ICAN είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα διεπιστώσαμε ένα πρόβλημα που το συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν τα λέμε dot wine ή dot vino ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να βρούμε κάποιες διεθνείς λύσεις για το θέμα του copyright το θέμα της προέλευσης, το θέμα της κληρονομιάς Νομίζω ότι αυτό είναι καλό να υπάρχει σε ουδέτερο επίπεδο και όχι να είμαστε προσκολλημένοι στι ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια το φόρουμ της διακυβέρνησης του δικτύου γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν έτσι κάπως ε, ε, σε πολύ πρωτόγονη φάση και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχουν προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ρούμπιχ. Εγώ πήγα εκεί ως εκπρόσωπος της ΣΤΟΑ. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό έχουμε με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δω τι είδου εναλλακτικέ λύσεις θα υπάρχουν στο μέλλον, τι πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη μας. Αυτό το φόρουμ της διακυβέρνησης διαδικτύου, το οποίο όπως σας είπα ε, παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο ρυθμιστικό ή συνένεσης γενικότερα με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει η ITU και πάλι από την άλλη πλευρά ο Ευρωπαίος Νομοθέτης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε πού βρίσκονται ποιες αρμοδιότητες. Ως ε, άμεσα ενδιαφερόμενος που μπορεί κανείς συμμετάσχει σε, μια παγκόσμια συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ο καθοριστικός ρόλος στο IGF ε, για να τον επιτύχει κανείς θα πρέπει να εξοικειωθεί λιγάκι με θέματα διακυβέρνησης και να δει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούμε και πρέπει να παίξουμε πρωτοποριακό ρόλο σε θέματα νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά ε, τα κανονιστικά Ινστιτούτα, τι μπορεί να επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή δεύτερον, τι είδους τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να προωθήσουμε, ε, να ε, προωθήσουμε νέες προδιαγραφές, να επιτύχουμε μια νέα αγορά με την απόλυτη εναρμόνιση. Υπάρχει και το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης. Ε, δεν είναι και το καλύτερο, δεν βοηθάει στο να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση. Για μας αυτό που ενδιαφέρει είναι να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς γίνεται με τις ε, γενικές ε, προϋποθέσεις που πρέπει κανείς να υπογράψει γενικούς όρους ότι συμφωνεί όταν κατεβάζει την έψα και η διαλειτουργικότητα της ΕΠΣΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και επίσης, ποιος έχει πρόσβαση στις συσκευές μας. Από ό,τι φαίνεται, εμείς ε, δεν είμαστε οι κυρίαρχοι και οι διοκτήτες ε, των ε, συσκευών μας, αλλά τρίτοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις συσκευές μας. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πραγματική πρόκληση σε σχέση με τα θέματα της ιδιωτικής σφαίρας. Γιατί αν μπορεί ο καθένας να ανοίγει την κάμερα ή να ανοίγει το μικρόφωνο το δικό μας και να παίρνει δεδομένα από τον υπολογιστή μας ή και να προσθέκει δεδομένα και ε, απλά πατάν, πατώντας ένα μικρό κουμπί ότι δέχεται κάποιους γενικούς όρους, αυτό νομίζω δεν είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να διερωτηθούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί νομίζω ότι στο μέλλον αυτό θα είναι ένα από τα κέρια θέματα. Πολύ σας ευχαριστούμε. Από το Κοινοβούλιο, όχι μόνο, από την Επιτροπή Ήτρε που ήρθατε και υποβάλλατε αυτή την αναφορά. Υποθέτουμε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το φόρουμ και η επόμενη συνεδρίασή του θα γίνει το Νοέμβριο του 2015 στη Βραζιλία. Και κάθε επιτροπή ζήτησε να στείλει αντιπροσωπεία σε ένα χρόνο από τώρα στη Βραζιλία για την ετήσια διάσκεψη του διαδικτυακού φόρουμου. Έσω έτοιμοι, συνάδελφοι. IGF, Βραζιλία. Επίσης, να προετοιμαστείτε για την επόμενη δική μας συνεδρίαση, στις 3 Δεκεμβρίου, πρωί-απόγευμα. Και 4, επίσης πρωί-απόγευμα. Σε 4 επεισόδια. Πάρα πολύ μεγάλη συνεδρία. Τα καλύτερα σας εύχομαι για τις επόμενες ημέρες και τα λέμε στο Στράσβουργο.